Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Äh, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη συνεδρίαση συγκρότηση σε σώμα. Είναι η πρώτη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Γεωργίας της νέας 1924. Ε, Έχουμε μερικά τυπικά θέματα να διεκπαιρεώσουμε πριν μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία. Πρώτα απ' όλα, έγκριση της ημέρης της διάταξης. Εάν δεν ε, υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνεται η ημέρης διάταξη όπως ε, προτείνεται. Α, η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και είναι η πρώτη μας συνεδρίαση και είναι η πρώτη φορά που απεβίωσε μέλος Επιτροπής μας ο κύριος Αντρέ Διονύσιο Μπράτφορτ να στείλουμε ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα ή επιστολή εκ μέρους Επιτροπής στην οικογένειά του. Πρόκειται για ένα συνάδελφο, σύντροφο της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών από τις Αζόρες ε, θα ήταν κανονικά μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και που απεβίωσε πριν από λίγες μέρες. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγγιλέρα. Βεβαίω, είναι στη μέση διάταξη ότι θα αναφερθούμε σε δύο λεπτά. Προβλέπετε. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα λοιπόν θέματα, να σας ενημερώσω για κάποια θέματα. Πρώτον, στη σημερινή μας συνεδρίαση ε, έχουμε κάλυψη από το ίντερνετ, ζωντανή, διερμηνία. Έχουμε όλες τις γλώσσες, εκτός από εστονικά, λετονικά, μαλτέζικα και γοηδελικά, Ερλανδικά. Όλες οι άλλες ε, προβλέπονται. Επίσης, υπάρχει ένα ε, πακέτο καλωσορίσματος για τα μέλη, όπου θα βρείτε κάποια λόγια καλωσορίσματος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΆΙΠΟΛ και ένα κατάλογο επαφών της Γραμματείας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την Επιτροπή Γεωργίας και για τις δραστηριότητες της περίοδου 2014-2019. Ίσως να σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα του δυστυχώς αποβιώσαντος ε, Άντρε Γιώργη Μπράτφορντ. Ο συνάδελφος ε, Αμάρο ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συνάδελφο ε, του Αντρέα Μπράτφορντ, παρόλο που ανήκουμε σε διαφορετικέ πολιτικέ παρατάξει στην Πορτογαλία, αλλά το γνώρισα και στην προεκλογική μα εκστρατεία συζητήσαμε για σημαντικέ πτυχέ τη κοινή ε, γεωργική πολιτική. Μάλιστα καταγόταν από μια εξόχω απόκεντρη περιοχή ε, και γι' αυτό ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Και με μεγάλη θλίψη, συντριβή, θα ήθελα να εκφράσω την ελληνική μου και την συμπαράστασή μου στην οικογένειά του. Και όπως είπε και η συνάδελφος, θα μπορούσαμε και εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας να στείλουμε είτε στην οικογένειά του, είτε στο Πορτογαλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα τα ειλικρινέστατά μας συλληπιτήρια για το χαμό του συναδέλφου Μπράτφορντ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Αμάρου. που αναφερθήκατε στο Σάνθο Bradford. Σας παρακαλώ να σηκωθείτε για να έχουμε ενός λεπτού Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Να περάσουμε τώρα στα επόμενα θέματα μέσα τη διάταξης. Εκλογή τρίτου αντιπροέδρου ή τρίτης αντιπροέδρου. Και η κυρία Αγγιλέρα. η κυρία Αγγιλάρ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο αυτές τις στιγμέ. Είναι σημαντικό να ανασκουμποθούμε και να ξεκινήσουμε αμέσως τη δουλειά μας. Και γι' αυτό είμαι εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, για το καλό των ε, Ισπανών και Ευρωπαίων αγροτών. Θα πρέπει λοιπόν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να ολοκληρώσουμε τι αρχαιρεσίε και την εκλογή των αντιπροέδρων. Τεράστια είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία με τη σύναψη τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Κανονικά δεν θα πρέπει να ψηφίζουμε, αλλά να υποβάλουμε προτάσει και να ακούμε κυρίω του ε, γεωργού και κτηνοτρόφου μα. Γι' αυτό κυρίε και κύριοι, συνεχίζει στα γαλλικά, κύριε Αγγιλάρ. Θέλουμε άμεση λύση. Και ε, σας ευχαριστώ που ε, μου επιτρέπετε να υποβάλω την υποψηφιότητα για την τρίτη αντιπροεδρία τη Επιτροπή, γιατί στόχο μα είναι να προσπίσουμε τα συμφέροντα όλων των αγροτών τη ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλάρ. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Πριν εκλέξουμε, κύριο Σουντεκάστρο. Ναι κύριε Πρόεδρε, εγώ εξ ονόματος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητα της κυρίας Κλάρα Αγγιλέρα ως Αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Μάκιντάρ. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, ε, κατανέμε τις ε, θέσεις των αντιπροέδρων με βάση το σύστημα DEONT. Και οι πρόεδροι των ε, επιτροπών συμφώνησαν με τις ε, πολιτικές ομάδες να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα, τον κανόνα ΔΕΟΝΤ. Το ίδιο ισχύει και για τι θέσεις των αντιπρόεδρων. Αν πιστεύετε λοιπόν σε αυτό το σύστημα και το στηρίζετε, όπως κάνουν πολλές πολιτικές ομάδες, κανονικά και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες προσυπογράφουν αυτό το κανόνα, και με βάση τον κανόνα ΔΕΟΝΤ, η θέση της τρίτης, του τρίτου αντιπροέδρου ανήκει στο ECR, στους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω εγώ την υποψηφιότητα της κυρίας Αγγιλάρ για τη θέση της τρίτης αντιπροέδρου της Επιτροπής Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κάνουμε τώρα την εκλογή, καταρχά, πώς υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Όχι. Οπότε να σας πω κάποια διαδικαστικά για να ξέρετε ακριβώς πώς γίνεται η εκλογή. Η κυρία Αγγιλέρα θέλει πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εγώ ασχολούμαι, για όσους το ξέρουν, για δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία στην Επιτροπή Γεωργίας και φυσικά προασπίζω τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Γεωργών και Κτηνοτρόφων και των Ευρωπαίων και των Ισπανών. Και γι' αυτό θα ήθελα να είμαι υποψήφια για τη θέση της Αντιπροέδρου. Φυσικά, φυσικά, οι συνάδελφοι θα αποφασίσουν αν θα με ψηφίσουν ή όχι. Αλλά δεν θα ήθελα να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικό με την άλλη υποψήφια, την κυρία Γκυλάρ. Αλλά ε, κρίνουμε σκόπιμο στους σοσιαλιστές να έχουμε και δικό μας υποψήφιο στο Προεδρείο στη θέση της τρίτης αντιπροέδρου. Γι' αυτό και είμαι υποψήφια της ομάδας μου για τη θέση αυτή της τρίτης αντιπροέδρου της Επιτροπής Άγκρη. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, τώρα κάποια διαδικαστικά θα τα διαβάσω στα αγγλικά. Για να ξέρετε ακριβώς πώς έχει η διαδικασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουμε το Προεδρείο της Επιτροπής Άγκρη και θα έχουμε τις χωριστές εκλογές ε, του ή της ε, τρίτου και τετάρτου αντιπροσώπου. Μπορεί να χρειαστεί να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά σήμερα. Λοιπόν, σας παρακαλώ και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να ελέγξετε ότι έχετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας. Είναι κανείς που δεν την έχει επάνω του. Α, εσείς, Χέντβικη. Is from the... Μήπως υπάρχει κάποιος αναπληρωτής από το ΕΛΚΑ που μπορεί να αντικαταστήσει τον κύριο Χέντβικη. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Οπότε είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Να ελέγξουμε αν λειτουργεί σωστά η ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα ελέγξουμε και ότι έχετε τις κάρτες σας. Okay, also wir haben... Λοιπόν, λοιπόν. 48 κάρτε είδαμε. 48. Πρέπει να ψηφίσετε όλοι. Δεν έχει καμία σημασία τι χρώμα, πράσινο, κόκκινο, άσπρο. Ψηφίστε όμως. Τώρα έχουμε ένα παραπάνω. Α, όχι, τώρα είναι 48. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 42, 43. Σας παρακαλώ. Πατήστε ένα κουμπί. Ένας συνάδελφος. Ένας μη γεγραμμένος παραπάνω. Α, εγώ δεν ψήφισα, ναι, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, έχουμε έναν μία εγγεγραμμένο παραπάνω. Α, τώρα είμαστε εντάξει. 48 παρόντες, 48 εψήφισαν. Α, πάλι ένας παραπάνω. Οι μη εγγεγραμμένοι μπορούν να καθαρίσουν, να ξεκαθαρίζουν ποιος ψηφίζει και ποιος όχι. Σας παρακαλώ βγάλτε την κάρτα ένας. Οκ. Okay. Άρεστα. Πέρας. Ωραία. Τώρα είμαστε λοιπόν σε θέση να ψηφίσουμε Λοιπόν, οι δύο υποψήφιες έχουν σχεδόν το ίδιο όνομα βέβαια. Αυτό είναι δυσχέρεια. Μπορεί να μπερδευτεί κανείς. Οπότε, προτείνω. Η κυρία Αγγιλάρα από το ECR είναι το πράσινο κουμπί. Η κυρία Αγγιλέρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες είναι στο κόκκινο κουμπί. Κόκκινο κουμπί. Λοιπόν, Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αγγιλάρ, πράσινο, Αγγιλέρα, κόκκινο. Ωραία, πέρας. Και η συνάδελφος Αγγιλάρ εκλέγεται με 27 ψήφους. Με 20 και 20 η κυρία Αγγιλέρα και μία ε, αποχή συγχαρητήρια. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στην εκλογή του ή της τέταρτου αντιπροέδρου. Υπάρχουν προτάσεις, η κυρία Μίλα. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνω τη συνάδελφο Έλση Κατάινεν. Είναι δεύτερη θητεία της τεταρτου διπροέδρου υπαρχουν προτασεις κυρια μιλα ευχαριστω πολυ προτεινω τη συναδελφο ελση καταινεν ειναι δευτερη θητεια της εδω στην ε, Επιτροπή Γεωργίας και θα χαρούμε αν την στηρίξετε. Έχουμε άλλες υποψηφιότητες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία θα ήθελα να α, καταθέσω την υποψηφιότητα της συναδέλφου Μπαξέτ Πυρμπακάς. Vielen Wir haben zwei... Ε, ωραία, έχουμε δύο υποψηφιότητες. Την κυρία Κατάινεν και την κυρία Πυρμπάκα. Ε, ε, υπάρχουν άλλε υποψηφιότητες. Α, η κυρία Πυρμπάκα. Ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτέ. Είμαι υποψήφια για τη θέση τη τέταρτη αντιπρόεδρου τη Επιτροπή Γεωργία. Η Γεωργία δεν είναι απλώ τομέα ε, στο οποίο βρίσκομαι τυχαία ε, και στην Επιτροπή αυτή ω μέλο. Εγώ είμαι ίδια Γεωργό και είναι ένα τομέα που ε, εξασφαλίζει βιοπορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Από έξι χρονών ασχολήθηκα με τους γονείς μου, με τη γεωργική μας εκμετάλλευση, και δίνω με του συνδικαλιστέ γεωργούς μάχη για να προστατεύσω τη γεωργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω των από απόκεντρων περιοχών. Δεν με ενδιαφέρουν οι κομματικές συγκρούσεις. Θέλω με ευφυα να συνεργαστούμε με όλου και να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Ανέκαθεν αυτό ήταν το ζητούμενο για μένα. Α είμαστε λοιπόν ρεαλιστέ και α προ... υπερασπίσουμε από κοινού την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Είμαι κυρίω μια συνδικαλίστρια που εξελέγει Ευρωβουλευτή σε ένα πολιτικό κόμμα. Σα ζητώ να με ψηφίσετε, γιατί είμαι γυναίκα, γεωργό, από εξόχω απόκεντρη περιοχή κατάγομαι. Και μάλιστα τα υπερπόντια διαμερίσματα αποκαλούνται εξόχω απόκεντρε περιοχέ ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 359 τη Ηθίκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να εκφράσω την, ε, την ευχή η ιδέα της διαφορετικότητας και της ισότητας ανδρών και γυναικών να μην είναι μια εξόχως απόκεντρη ιδέα για την Επιτροπή Γεωργίας. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Περμπάκας. Η κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο και να ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο ε, στην, που, ασκούμε, που επιτελούμε στην Επιτροπή Γεωργίας. Είμαι για δεύτερη συναπτή κοινοβουλευτική θητεία Ευρωβουλευτής και επίσης μέλος της Επιτροπής Γεωργίας για δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία μελέτησα, σπούδασα και δίδαξα στα θέματα της γεωργίας και των φυσικών πόρων. Ήμουν για 11 χρόνια και εθνική βουλευτής και η προάσπιση της παραγωγής τροφίμων και γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μου δημιουργεί μεγάλη, μεγάλο ενθουσιασμό και θέλω να προωθήσω αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κυρία Κατάιν. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Και αυτή τη φορά έχουμε δύο υποψήφιες θα εκλεγεί λοιπόν η υποψήφια που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψήφων. Οπότε, λοιπόν, πάρτε τις κάρτες σας. Πράσινο είναι η κυρία Κατάιναν και κόκκινο η κυρία Πυρμπάκας. Λοιπόν, άρχεται. Λοιπόν, λέμε πράσινο και πάλι επαναλαμβάνω. Πράσινο, έναν, κόκκινο, Πιερ Μπάκα. Πέρα προφορία. Εξελέγει η κυρία Κατά έναν. 29 ε, με ψήφου πήρε η κυρία Κατά 9 η κυρία Πυρμπάκα και ε, υπήρξαν και 9 αποχέ. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann können wir... Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της τη διάταξη. Όμω πρέπει να περιμένουμε γιατί δεν έχει έρθει ο επίτροπο. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε τον Επίτροπο, οπότε σύντομη διακοπή. Σας παρακαλώ. Καλύτερα μην σηκωθείτε καν, γιατί μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή ο Επίτροπος να μην χάσουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, σα παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε χωρί άλλη καθυστέρηση και να καλωσορίσω θερμά τον Επίτροπο για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Φιλ Χόγκαν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Πολύ καλό είναι στην αρχή μιας νέα θητεία να επιδιώκουμε το διάλογο με τον Επίτροπό μα, τον Επίτροπο Γεωργία. Και είναι σαφές ότι έχουμε μπροστά μας πολλά σημαντικά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, είναι στην ημερήσια διάταξη οπότε μια συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη. Μια συζήτηση όπως αυτή που θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα μαζί σας Πρώτα απ' όλα έχουμε την πρόταση για την μεταρρύθμιση της ε, γεωργικής πολιτικής. Τρεις διαφορετικοί κανονισμοί και οι επιπτώσεις της ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με το Mercosur στην ε, γεωργία της Ένωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμφωνία που επετεύχθη μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεις στις 28 Ιουνίου. Και αν μας το επιτρέπει ο χρόνος, θα δούμε και τις επιπτώσεις για τη Γεωργία της ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου που υπεγράφει στις 30 Ιουνίου με το Βιετνάμ. Θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και θα δούμε και τα πορίσματα της ομάδας υψηλού επίπεδου για τη ζάχαρη. Κύριε Επίτροπε, σας δίνω το λόγο Ίσως για τους νέους συναδέλφους, πριν δώσω το λόγο για τον Επίτροπο, διαδικαστικά, ο Επίτροπος θα κάνει την αρχική του ομιλία. Κατόπιν θα πάρουν το λόγο οι 7 συντονιστές, ο καθένας δύο λεπτά. Και το λέω εξ αρχής, αγαπητοί συνάδελφοι, προτίθεμε να ε, επιβάλλω την τήρηση του χρόνου. Μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος και μετά θα πάρουν το λόγο οι επόμενοι συνάδελφοι. Ένα λεπτό καθένας. Κύριε Επίτροπε, σας δίνω το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Λίντς, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ εδώ σήμερα το απόγευμα και να μπορέσουμε να συζητήσουμε αμέσως μετά τη σύστασή σας σε σώμα στην Επιτροπή Γεωργίας και να σας συγχαρώ καταρχάς όλους για την πρόσφατη εκλογή ή επανεκλογή σας και θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω συγχαρώ εσάς κύριε Πρόεδρε και τους αντιπροέδρους της Επιτροπής και τους συντονιστές ε, της κάθε πολιτικής ομάδας. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας για το κοινό συμφέρον των γεωργών μας. Καταρχάς ε, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω την ε, ε, αλληλεγγύη μου και την, ε, τα συλλεπιτήριά μου για το χαμό του συναδέλφου σας, του κυρίου Μπράτφορντ, ο οποίος απεβίωσε προσφάτως. Δεν το γνώριζα, ήταν μέλος της Επιτροπής σας, αλλά αναγνωρίζω ότι ήταν μεγάλη απώλεια για την οικογένεια και τους φίλους τους να έρθει κάποιος εδώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αποβιώσει τόσο σύντομα μετά την εκλογή του. Βλέπω πολλές ε, νέες φυσιογνωμίες, αλλά και πολλές οικίες φυσιογνωμίες εδώ. Ε, φαίνεται ότι εδώ μπροστά έχουμε τις συνηθισμένες φυσιογνωμίες. Ε, χαίρομαι που βλέπω ένα πολύ καλό αμάλγαμα νέων και πιο έμπειρων ευρωβουλευτών. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή αυτή συνέβαλε ουσιαστικά σε πολλά θέματα. Ξεκινήσαμε με το ρωσικό εμπάργο και χρειάστηκε να ασχοληθούμε και με τις συνέπειες του εμπάργου, ε, την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης και βλέπω και τον προκάτοχό μου, τον κύριο Τσόλος εδώ. Είχαμε τον κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα, ο κύριο Χάουσλινγκ και η Σκιώδη, ε, τον κανονισμό Omnibus με τον κύριο Ντεκάστρο και τον κύριο Ντε και την οδηγία για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικές. Ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα, του οποίου ηγήθηκε ο κύριο Ντεκάστρο και φυσικά οι Σκιώδη διδερμάτισαν και πολύ σημαντικό ρόλο για τα συμπεράσματα για αυτή ε, τα πολύ σημαντικά θέματα και μέσω των εργασιών αυτή τη επιτροπή καταφέραμε να κάνουμε τη ζωή των γεωργών μας ε, και των διοικήσεων κατά την άποψή μου καλύτερη και πιο εύκολη για πολλά ε, και ακαθόδη γεωργικά θέματα που ε, μπορεί να ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα. Η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, για παράδειγμα, για πρώτη φορά εισήχθη ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για προστασία κατά των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, για να υπάρχει μια καλύτερη αλυσίδα ε, διανομής τροφίμων, το οποίο αφορά και την ίδια την επιβίωση των γεωργών μας σε κάποιες περιπτώσεις. Όπω είπα κύριε Πρόεδρε λοιπόν, δεν μπορώ να καλύψω κάθε θέμα σήμερα, αλλά προσβλέπω στι ερωτήσει σα, και θα ήθελα να καλύψω κάποια επίκαιρα ζητήματα στον κόσμο της γεωργίας και όσα απασχολούν φυσικά τους γεωργού μα αυτή τη στιγμή. Ε, σήμερα ε, έχουμε οικονομική και περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική και η γεωργία λοιπόν είναι κεντρικός μοχλός ε, του αγροδιατροφικού τομέα, παρέχει άμεσα και έμεσα δουλειές για 44 εκατομμύρια ανθρώπων οι εξαγωγές ε, αγροδιατροφικών προϊόντων ήταν πάνω από 147 ε, δις ευρώ, που σημαίνει πλεόνασμα περίπου 22 δις ευρώ. Άρα η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει πάρα πολύ στην προστασία των φυσικών μας πόρων, το έδαφος, ε, το νερό, τη βιοπικιλότητα και το 57% της γης μας, 85% αν προσθέσουμε και τις δασικές εκτάσεις και φυσικά μας ζητάτε να κάνουμε περισσότερα στις νέες προτάσεις για την νέα ΚΑΠ. Η πολιτική υποστηρίζει φυσικά και τις περιοχές της Υπέθρου που είναι περίπου ε, η κατοικία του ε, μισού πληθυσμού των Ευρωπαίων και παρέχει τη βιοπικιλότητα. Η πολιτική του μέλλον θα πρέπει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ε, ε διατήρηση του περιβάλλοντος και φυσικά αυτό αφορά και την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα ενώπιον κινδύνων και κρίσεων και φυσικά το να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρεται από τις νέες τεχνολογίες και την ολοκλήρωση της έρευνας και της τεχνολογίας για διάφορες γεωργικές πρακτικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τη νέα γενιά των γεωργών, τους νέους μας ανθρώπους εδώ. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε περαιτέρω και την εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικών ε, θεμάτων στη γεωργία. Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υδάτων, να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα, να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και ου μόνο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και θέματα που αφορούν ε, τη δυνατότητά μας να εξασφαλίσουμε ότι θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες παραγωγής τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια. Στις προτήσεις για την ΚΑΠ συζητούμε επίσης και το θεματολόγιο για την ε, υγιή ζωή ε, και θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων, το επίπεδο των φυτοφαρμάκων, αντιβιωτικά κλπ. Η γεωργία λοιπόν θα πρέπει να είναι τμήμα της λύσης και η γεωργία θα πρέπει να είναι τμήμα της λύσης, αλλά το 2019 έως 2024 στο στρατηγικό σωματολόγιο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν επίσης στα τέλη Ιουνίου ότι πρέπει να υπάρχει και μια Ευρώπη η οποία θα είναι ουδέτερος προς το κλίμα, πράσινη, δίκαιη και κοινωνική. Η νεοκλογήσα πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Βαντερ αναφέρθηκε στην έκθεση ε, σε κλιματικές συνθήκες για τους γεωργούς και αναφέρθηκε σε, μια, σε ένα New Deal για τους ε, ε, γεωργούς. Η γεωργία λοιπόν θα πρέπει να είναι έτοιμη για να συμβάλλει και αυτή σε αυτό τον εμβληματικό στόχο. Η ΚΑΠ επίση θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι προστατεύουμε και τις περιοχές της υπαίθρου, δημιουργώντας θέσει εργασίας και ανάπτυξη και να προσφέρουμε και μια προοπτική στις κοινότητε της υπαίθρου και να αντιμετωπίζουμε και τις άμεσες κοινωνικές ανάγκες τους. Όσον αφορά το σεβασμό, το ε, Συγγνώμη, όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία πρόταση και επειδή είναι πολύ γνωστές οι συνθήκες ε, ε, βάσει των οποίων έγιναν, κυρίως το Brexit, μένω της άποψης ότι είναι μία καλή αρχική θέση και είναι και μία θέση η οποία θα εξασφαλίσει ότι η ΚΑΠ θα διαδραματίζει πλήρη ρόλο στην προστασία των γεωργών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ε, έχουν ε, οι γεωργοί. Το 26% του προϋπολογισμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να παραμείνει στη γεωργία. Το 96. Επομένως, προτείνουμε 365 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 δις επιπλέον δίνονται για έρευνα και ανάπτυξη στις ε, γεωργικές και περιοχές και περιοχές της υπαίθρου και θέλουμε να υποστηρίξουμε και τον εξυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ξέρω ότι πολλοί από εσά θα εκφράσουν και την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση για την ΚΑΠ. Επομένως, προσβλέπω στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, τώρα πλέον τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει να δεχτούν ή να τροποποιήσουν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν υπάρχει πρόταση να αυξηθεί η χρηματοδότηση τη ΚΑΠ. Ε, φυσικά αυτή η πρόταση θα έρθει από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ ευχαρίστω να το δεχτεί η Προεδρία της Φιλανδίας έχει δώσει ως προτεραιότητα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο πρόγραμμά της. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο, διότι θα είναι δύσκολη δουλειά, αλλά θα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος, να δώσουμε ασφάλεια και προβλεψιμότητα για τους γεωργούς ε, και υπάρχουν και αποφάσεις που ξέρω ότι πολλοί από αυτούς ε, περιμένουν ε, και γι' αυτό και η προβλεψιμότητα είναι πολύ σημαντική. Ελπίζουμε λοιπόν να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του έτους. Κύριε Πρόεδρε, πριν από τις ευρωεκλογέ, η Επιτροπή σας ε, ψήφισε για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική ΚΑΠ. Ξέρω ότι τα συζητάτε εδώ όσον αφορά το τι μέλη γενέστε και εγώ δεν θα εμπλακώ φυσικά σε αυτή τη συζήτηση, αλλά ελπίζω να αποφασίσετε να συνεχίσετε τα όσα έχουν ήδη γίνει και ε, υπάρχει πολύ καλή δουλειά που έγινε από τους τρεις εισηγητές όσον αφορά την προετοιμασία της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμείς αιτιολογήσαμε το 96% του προηγούμενου προϋπολογισμού να παραμείνει στη Γεωργία και είπαμε ότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε την πολιτική. Υπάρχουν συγκεκριμένα ε, σχέδια για να αυξηθεί και το επίπεδο φιλοδοξίας για το περιβάλλον και το κλίμα. Όταν λοιπόν θα φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο του Πολιτικού δημοσιονομικού ε, πλαισίου, ελπίζουμε εντός του έτους, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα θέλουν να ξέρουν για ποιο λόγο η Επιτροπή σας ή και άλλες επιτροπές ε, ζητούν περαιτέρω αύξηση στον προπολογισμό, ακόμα και για τον προπολογισμό της ΚΑΠ. Και πού θα δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή σας να μπορέσει να αποδείξει σε όσους βρίσκονται γύρω από το τραπέζι όταν ψάχνουν για περισσότερα χρήματα ότι μπορείτε να εξηγήσετε για ποιο λόγο ζητάτε περισσότερα χρήματα. Εάν και εφόσον το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβουν θέση όσον αφορά την πρόταση για το 2020, μπορούμε να περάσουμε ε, και στα υπόλοιπα. Και μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετέχει στον τριμερή διάλογο με ανοιχτή ε, προσέγγιση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Όπω γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών Μερκοσούν, Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, επετέφθη εχθέ μετά από 20 ακριβώ χρόνια διαπραγματεύσεων. Είμαι ικανοποιημένο διότι η συμφωνία είναι ισορροπημένη, αλλά επίση και πλήρη και φιλόδοξη. Και δέχομαι πλήρω ότι αποτελεί πρόκληση για κάποιου γεωργικού τομεί. Ωστόσο, έχουμε εξασφαλίσει και πολύ σημαντικές ευκαιρίες για κάποιους τομείς της γεωργίας. Τον νίνο, τα ενοπνευματώδη ποτά, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, μεταποιημένα προϊόντα, για να σας πω κάποια εξ αυτών και μετά από πολύ σημαντικές εμπορικές συμφωνίες όπως αυτή της Ιαπωνίας, του Μεξικού και του Βιετνάμ που ε, όλες αυτές έχουν προσφέρει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους ε, γεωργούς και παραγωγούς ήμασταν σε σημαντική στάση όσον αφορά το Μερκοσούρ και εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ο όρο Μερκοσούρ δημιουργούσε συγκεκριμένη εικόνα στην Γεωργία που δεν ήταν ε, πάντα θετική. Ο στόχο όπω γίνεται με τι διαπραγματεύσει είναι να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να μειώσουμε τι προκλήσει. Ε, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να προσπαθήσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τη Γεωργία, ενώ ταυτόχρονα προώθησε και άλλα συμφέροντα. Αυτά λοιπόν τα συμφέροντα εξασφαλίζονται μέσω τη εντολή που έδωσαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολύ σημαντικά προϊόντα, όπω για παράδειγμα το βόηο κρέα, ε, τη ζάχαρη, ε, και να υπάρχουν ε, περιορισμένοι δασμοί εισαγωγή, ε, ποσοστώσεις, περιοχές και δικλείδε ασφαλείας για κάποια από τα πιο ευαίσθητα προϊόντα μας και, εάν χρειαστεί, ακόμα και μία δέσμη χρηματοοικονομικής στήριξη. Η Επιτροπή μας θα πρέπει τελικά και το Κοινοβούλιο φυσικά να καταλήξει συμπεράσματα για το ποιες προκλήσεις προκύπτουν από αυτό. 4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αξία αυτής της συμφωνίες για τους εξαγωγούς και αγροτροφικών προϊόντων. 345 γεωγραφικές ενδείξεις έχουμε προσπίσει με τη συμφωνία αυτή. Πολύ θετική έκβαση για τους παραγωγούς ε, προϊόντων υψηλής ποιότητας. Και δεν άκουσα τίποτα για τα 339 ονόματα που έχουν τύχει προστασία και που είναι ευρωπαϊκά. Το επίπεδο προστασία που επιτύχαμε είναι το ίδιο που υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μερικές λίγες εξαιρεσει που περιορίζονται σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και ε, λόγω της απόστασης. Φυσικά ε, για το βόλιο, ε, τα πουλερικά και τη ζάχαρη, που είναι τα βασικά προϊόντα, τα εξασφαλίσαμε. Θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χορηγηθεί περιορισμένα και με πολύ αυστηρούς ελέγχους στις χώρες Μερκοσούρ και λαμβάνει υπόψη η πρόσβαση αυτή τις ανησυχίες των ε, Ευρωπαίων Γεωργών. Και μάλιστα θα έχουμε σταδιακή εφαρμογή των ποσοστώσεων και μάλιστα σε έξι ετήσιες φάσεις που θα είναι ίσες. Και εκτός από τις ε, ποσοστώσεις της δασμολογικές που θα προστατεύσουν ευαίσθητους τομείς, έχουμε στη Συμφωνία έναν ε, διμερή μηχανισμό ασφαλιστικής δικλίδας προκειμένου να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά μέτρα για να ρυθμίσει τις εισαγωγές σε περίπτωση απροσδόκητης και σημαντικής αύξησης των ε, εισαγωγών που ε, προκαλεί, απειλεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στις, στις ε, εσωτερικές αγορές. Και αυτό καλύπτει και τα γεωρικά προϊόντα που εμπίπτουν στι δασολογικές ποσοστώσεις και για πρώτη φορά καταφέραμε να συμπεριλάβουμε μια τέτοια ρήτρα σε Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Μέχρι στιγμής έχει ισχύσει μόνο για τομείς που ήταν απόλυτο απελευθερωμένοι. Και ένα σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι εξασφαλίσαμε οι δασμολογικές αυτές ποσοστώσεις να, να τις διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με εισαγωγικέ άδειε. Έτσι εμεί θα ελέγχουμε τη ροή αγαθών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία αυτής της πτυχής της συμφωνίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε ένα δισεκατομμύριο ευρώ ενίσχυση αποκλειστικά του γεωργικού κλάδου σε περίπτωση που η εφαρμογή τη Συμφωνία θα δημιουργήσει τρευλώσει στην αγορά γεωργικών προϊόντων. Αυτή η επιπλέον χρηματοοικονομική στήριξη θα χρηματοδοτήσει μέτρα που υπήρχαν στα πλαίσια τη κοινή οργάνωση αγορών και όπω έχει δείξει πρόσφατη μα πείρα έχουμε τα απαραίτητα μέσα πολιτική στην κοινή γεωργική πολιτική για να παρέμβουμε αποτελεσματικά στην αγορά εφόσον το απαιτεί κάτι τέτοιο η κατάσταση και κάτι τέτοιο συνέβη ήδη το 2015 και 2016. Και μάλιστα ε, μόνο αποκλειστικά για το γεωρικό τομέα πρώτη φορά έχουμε τόσο σημαντική υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο κλάδο σε, στα πλαίσια μιας εμπορικής συμφωνίας. Αναφέρθηκε ότι με τη συμφωνία χαλαρώνουμε τα υγειονομικά μα πρότυπα και προδιαγραφέ. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το αντίθετο μάλιστα ισχύει με τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διατρανώνουμε την αρχή τη προφύλαξη με τη συμφωνία αυτή και δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις ε, αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κανόνες ασφάλειας. Όλα τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιμένοντας την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών μας των υγειονομικών ουσιαστικά βελτιώνουμε τις υγειονομικές προδιαγραφές και πρότυπα και στις χώρες Μερκοσούρ. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό το θέμα των υγειονομικών μας προτύπων και θα πρέπει να μείνουν όσα έχουν αυτά τα πρότυπα και προδιαγραφέ με πλήρη ελέγχου που γίνονται από τα κράτη-μέλη, που γίνονται και από τη δική σα πατρίδα κύριε Χόισλινγκ. Και υπάρχει μερικέ φορέ η ψευδέστηση, και δεν είναι η πρώτη φορά κύριε Χόισλινγκ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει χαμηλότερε προδιαγραφέ για τα εισαγόμενα προϊόντα από ό,τι ισχύει για τα τοπικά προϊόντα. Αυτή η ψευδέστηση οφείλεται σε παραπληροφόρηση και θα πρέπει να διορθωθεί. Για να δούμε τι γίνεται με τη Βραζιλία, για παράδειγμα. Μόνο μερικέ περιοχέ μπορούν να εξάγουν προϊόντα του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Βραζιλία. Και η βασική περιοχή παραγωγή βόλου κρέατο στη νότιο Βραζιλία απέχει πολύ από την περιοχή του Αμαζονίου. Και το λέω για όσου ξέρουν και τη γεωγραφία. Μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα λιγότερο από 1% των σφαγείων έχουν λάβει την έγκριση την ευρωπαϊκή για εξαγωγές. Και μάλιστα τα καλύτερα σφαγεία έχουν λάβει αυτή την άδεια και την έγκριση για να εξάγουν. Και μάλιστα υπάρχει ένα πάγωμα για την προσθήκη οποιοδήποτε ε, νέου σφαγίου στον κατάλογο με τα επιτρεπόμενα σφαγεία για τις εξαγωγές. Και μάλιστα θα πρέπει να γίνεται αποστέωση και ορίμανση όλων των παρτίδων. Και μάλιστα μόνο από ε, ελέγχους ε, και μετά από ε, έλεγχο των εγγράφων και της ταυτότητας και σωματικών ελέγχων επιτρέπεται ε, η πραγματοποίηση της εξαγωγής. Και μάλιστα, χάρη στις διατάξεις αυτές, ε, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για το Μερκοσούρ. Γιατί μερικές φορές γίνεται πολύ επιλεκτική αναφορά κάποιων στοιχείων. Βέβαια, αναφέρθηκαν οι ανησυχίες για την για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο τη συμφωνία. Ε, και φυσικά σίγουρα η συμφωνία θα πρέπει να γίνεται ει βάρο του περιβάλλοντο και του κλίματο. αντίθετα να προωθεί βιώσιμη ανάπτυξη. Και μάλιστα περιλαμβάνεται και διαδικασία επίλυσης διαφορών σε περίπτωση παραβίασης οποιοδήποτε πτυχή τη συμφωνία. Και το Μερκοσούρ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμευθεί ρητά να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Παρισίων και του στόχου τη. και συμφώνησαν να συνεργαστούν για τι περιβαλλοντικέ πτυχέ τη εμπορική συμφωνία. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της ε, αποψήλωσης των δασών και να σεβαστούν τις εθνικές ε, δεσμεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Για παράδειγμα, η εθνικά καθορισμένη ε, συνεισφορά της Βραζιλίας για τη Συμφωνία των Παρισιών εξασφαλίζει απόλυτη απαγόρευση της παράνομης υλοτομίας και μάλιστα έχει ανα, δεσμευθεί να αναδασώσει τεράστιες εκτάσεις μέχρι το 2020 και φυσικά να απαγορεύσει και να καταργήσει τις ε, μη βιώσιμες πρακτικές. Και αυτό δείχνει την αξία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και, της, και του ανοίγματο αγορών με εταίρους που σέβονται και τηρούν τις δικές μας προδιαγραφές και κανόνες. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να επικυρώσετε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συμφωνία, κάνοντα μια εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των πτυχών τη συμφωνία. Αλλά για να βοηθήσουμε τη διαδικασία αυτή τη αξιολόγηση. Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας είναι στη διάθεσή σας και θα σας ε, ενημερώνουμε τακτικά για, το, για την έκβαση και των, ε, των μελετών αντικτύπου που θα ισχύσουν και για αυτή τη συμφωνία αλλά και τις άλλες με τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Ιαπωνία που θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. Φυσικά μια τέτοια γενική επισκόπηση δεν ε, καλύπτει με μονομένες ανησυχίες. Χρειάζεται πιο ευρύτης ανάλυση και πιο ε, ενδελεχής εξέταση. Και θα, θα σας στείλουμε τα, τις μελέτες αντικτύπου για όλους τους επιμέρους τομείς. Σε περίπτωση που δεν προλάβω τώρα να απαντήσω στις ανησυχίες σας για πολύ πιο περίπλοκα και λεπτομεριακά θέματα, πολύ ευχαρίστω να σας παραπέμψω στις ε, υπηρεσίες μας για να σας απαντήσω λεπτομεριακά. Για το Βιετνάμ τώρα. Ε, συντομία, πρόσφατα έχει συναυθεί η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και η Συμφωνία Προστασία Επενδυτή μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περιεκτική και φιλόδοξη συμφωνία. Μάλιστα, ε, πρώτη φορά έχουμε τόσο φιλόδοξη συμφωνία με αναπτυσσόμενη χώρα. Ε, και η δεύτερη μετά τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Και γενικός μας στόχος είναι οι συμφωνίες να γίνονται μεταξύ περιφερειών, όπως τις περιοχές ΑΣΕΑΝ. Έτσι έχουμε πρόσβαση σε μια αγορά 90 εκατομμύριων, που είναι η αγορά του Βιετνάμ, προκειμένου να εδραιώσουμε την παρουσία, την παρουσία μας σε μια από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου. Και μάλιστα είναι θετική η, συνέ, η επίπτωση της συμφωνίας και στη Γεωργία, γιατί χάρη στην απελευθέρωση την εμπορική, άνοιξε μέσα, θα ανοίξει μέσα σε τρία χρόνια η αγορά Βορειοκορεάτου, σε δέκα χρόνια των πολερικών, ε, για την οπνευματώδη σε 7 χρόνια πλήρη απελευθέρωση, ενώ μέχρι στιγμή έχουμε δασμούς μέχρι και 25% για τους τομείς αυτούς. 3 ε, με 5 χρόνια θα απελευθερωθούν τα γαλακτοκομικά, 9 το χοιρινό κρέα, απορροκυπευτικά 3 με 5 χρόνια και πολλά άλλα προϊόντα γεωργικά ε, σε 5 με 7 χρόνια. Και στην περίπτωση αυτή με το Βιετνάμ καταφέραμε να προστατεύσουμε ευαίσθητους κλάδους, το ρύζι, το άμυλο, ε, την εθανόλη, τα αυγά, τα μανιτάρια και ούτω καθεξής. Και μάλιστα 159 ε, προϊόντα που καλύπτονται από γεωργικές ενδείξεις προστατεύονται από παραποίηση και από μίμηση. Και μάλιστα οι γεωργικές ενδείξεις ε, στο Βιετνάμ αφορούν ευρωπαϊκά προϊόντα από παραδοσιακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωση, κάτι που βοηθά τους Ευρωπαίους γεωργούς και τις μικρές επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου λοιπόν με το Βιετνάμ είναι πολύ θετική για τους παραγωγούς τροφίμων και τους αγρότες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αυξήσουν σε εξαγωγές τους προστατεύοντας, παράδειγμα, το παράλληλα το περιβάλλον. Και είναι από τις σημαντικές ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που ευνοεί τους παραγωγούς. Με ρωτήσατε και για τις συνομιλίες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Είναι πολύ έντονε οι διαπραγματεύσει που γίνονται στον ΠΟΕ αυτή τη στιγμή στη Γενέβα, γιατί υπάρχουν ε, όλο και περισσότερε ε, μονομερεί αποφάσει που γίνονται ειδικά στι σχέσει ε, Ηνωμένων Πολιτειών και κίνα. Και μάλιστα οι προσφυγέ που έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείε στο δευτεροβάθμιο σώμα του ΠΟΕ έχουν δυσχεράνει το σύστημα. Εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε την πολυμέρεια και όχι να τη διαλύσουμε. Και σε ό,τι αφορά τη γεωργία, τόνισα πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο και για τη γεωργία μα. Θέλουμε ένα πολυμερέ εμπορικό σύστημα που θα δράζεται σε αυστηρού κανόνε. Και αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τον ΠΟΕ ε, για να στηρίξουμε το μέλλον της γεωργίας. Γιατί βλέπουμε ήδη πόσο μονομερείς δράσεις μπορούν να παραβλάψουν ε, το εμπόριο. Αυτό συνέβη με την περίπτωση των επιτραπέζων ελιών από την Ισπανία. Προσπαθούμε λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο στα θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ε, στα θέματα της αλίας και στα θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Βέβαια, πολλά θέματα είναι συναφή με την πρόοδο που γίνεται στη Γεωργία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι γεωργικές επιδοτήσει. Θα πρέπει λοιπόν τι συνομιλίε αυτές να τις ε, θεωρήσουμε ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. Και εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τον ΠΟΕ. Και ε, οι η περισσότερη υποστήριξη είναι για το πράσινο κουτί που δεν αφορά τη γεωργία. Και θα συνεχίσουμε ε, να προωθούμε τις συζητήσεις. Και θα πρέπει να περιοριστούν τα μονομερή μέτρα Κίνας, Ινδίας ε, και ε, Ηνωμένων Πολιτειών που πρόσφατα ενέκρινε πακέτο 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγροτικών ενισχύσεων θα πρέπει ο πολυμερής μηχανισμός που μέχρι τώρα λειτουργούσε να συνεχίσει να λειτουργεί. Χωρίς όμως μεταρρύθμιση άμεση, το σύστημα θα παραλύσει μέχρι τα, τέλος του τρέχο, τα τέλη του τρέχοντος έτους. Και μάλιστα στο δευτεροβάθμιο σώμα χρειάζονται, χρειάζεται τρεις ψήφοι και όχι μία. Και από την Υπουργική Διάσκεψη του Buenos Aires το Δεκέμβριο του 2017 δεν είχαμε καμία πρόοδο. Οπότε για την επόμενη πολιτική διάσκεψη του Ιουνίου του 2020, του 2020 δεν είναι ακόμη πολύ θετικές οι προοπτικέ. Αυτά κύριε Πρόεδρε, έβαλα τα δυνατά μου για να συνοψίσω τα πιο επίκαιρα θέματα στον σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου και ε, περιμένω τώρα τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε για τις ε, αναλυτικές σας ε, παρατηρήσεις και το ότι ασχοληθήκατε με όλα τα θέματα τα οποία ανέφερα. παρόλα αυτά έχω την εντύπωση, βλέποντας τα βλέμματα των συναδέλφων, ε, πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά για να πείσουμε όλους τους συναδέλφους. Λοιπόν, οι συντονιστές πρώτα απ' όλα. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε μια ομάδα σκεπτών του συναδέλφου Πάλλοντε Κάστρο. θέλω να τους καλωσορίσω. Μια ομάδα Οχτώ μελών του Προεδρικού Συμβουλίου της Ιταλικής ε, Συνομοσπονδίας ε, Γεωργών. Καλώς ήρθατε. Οπότε. Λοιπόν, οι συντονιστές. Ο Herbert Ντόρφμαν, πρώτος δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ε, ήρθατε, αξιότιμη κύριε Πίτροπε. Η ομάδα μου Χαίρετε που ήδη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας είστε εδώ για να ξεκινήσετε ή μάλλον να συνεχίσετε τον διάλογο που πάντα είχατε μαζί μας. Αναφερθήκατε σε μια σειρά από θέματα και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, μόνο δύο-τρία μπορώ να αναφέρω. Τα πιο σημαντικά θέματα τι επόμενε εβδομάδε και μήνε για μα εδώ στην Επιτροπή είναι σίγουρα πρώτα απ' όλα η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Όπω ξέρετε, κατά την προηγούμενη θητεία υπήρξαν πολλέ προτάσει και γι' αυτό λήθησαν αποφάσει από την Επιτροπή μα και εμεί από το ΕΛΚ θέλουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι αποφάσει ω βάση, αλλά να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης τις γνώμες των διαφόρων συναδέλφων και οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα πρέπει ε, να μας βρίσκουν όλους σύμφωνος για να μπορούμε να τις υποστηρίξουμε και έναντι των γεωργών μας. Νομίζω ότι θα βρούμε έναν ε, καλό τρόπο να συνεργαστούμε. Έχετε δίκιο. Η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι το πιο σημαντικό θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να πιστούν για να μην ε, λάβουν χώρα οι προταθήσεις περικοπές. Ξέρω ότι οι περικοπές προτάθηκαν ε, για το δεύτερο πυλώνα, την ανάπτυξη της υπαίθρου, θα οδηγήσουν σε τεράστια προβλήματα. Και βρίσκω πολύ θετικό κάτι που δεν έχει υπογραμμιστεί μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής, το Ταμείο για την ε, Έρευνα και την Ανάπτυξη των 10 ε, δισεκατομμύριων θα βοηθήσει να ε, έχει ένα βιώσιμο μέλλον η Γεωργία στην Ευρώπη. Για τη Μερκοσούρ, τη συμφωνία με το Μερκοσούρ, ε, νομίζω ότι υπάρχει λιγότερο ενθουσιασμό από το πώ το περιγράψατε. Πολλοί Γεωργοί ανησυχούν για τη συμφωνία αυτή, γιατί θίγει κάποιου ε, τομεί. Και κάτι ακόμη. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και το θέμα του Brexit, που επίκειται θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για την ε, αγορά γεωργικών προϊόντων. Είναι ένα σημαντικό θέμα που θα μας απασχολήσει του επόμενους μήνες και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω τον Επίτροπο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ αγαπητέ Επίτροπε Χόγκαν και σα ευχαριστώ και για το γεγονός ότι θυμήσατε στην εισαγωγή σας και πολύ σημαντικούς σταθμούς ε, που καταφέραμε εμείς εδώ στην Επιτροπή, όπως για παράδειγμα την οδηγία για τις αθέμητες πρακτικές και τον κανονισμό Omnibus. Όσον αφορά την ΚΑΠ, ε, σίγουρα η Επιτροπή μας θα πρέπει να δεσμευθεί και να ασχοληθεί με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον των γεωργών μας. Ένα θέμα ε, για το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αρκετέ επικρίσει. Δεν σα κρύβω ότι στην ομάδα μα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ονειρεύονται μια νέα νομοθετική πρόταση για την κοινή γεωργική πολιτική. Βεβαίω, ε, δεν θέλουμε να πετάξουμε στα σκουπίδια όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ε, τώρα, συγγνώμη, θα χρειαστεί όμως να σκεφτούμε κυρίως το θέμα του προϋπολογισμού, να εγκρίνουμε έγκριση ε, του ΣΚΑΠ όταν δεν έχουμε ιδέα για τον προπολογισμό. Δεν ξέρουμε τον Οκτώβριο θα υπάρξει Brexit ή όχι ε, και τι συνέπειες θα υπάρχουν για τον προπολογισμό από τον Brexit. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το Mercosur, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Ντόρφμαν. Υπάρχουν υπάρχουν και πολλές επικρίσεις. Ε, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καν καταλάβει και για ποιο λόγο επιταχύναμε στο τέλος της θητείας ε, ακόμα και γιατί δεν έχει γίνει συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια συζήτηση την οποία σίγουρα θα κάνουμε, θα κάνει εδώ η Επιτροπή μας ώστε να έχουμε και λίγο πιο σαφή εικόνα για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτή η συμφωνία για τους γεωργούς μας. Και τέλος, ε, κύριε Επίτροπε, δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα προλάβουμε να οργανώσουμε την μεταρρύθμιση μέχρι το 2020, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να παρουσιάσουμε μεταβατικό κανονισμό για να δώσουμε ε, και ασφάλεια στους γεωργούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Μίλλερ, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Και το γεγονό ότι υπερασπίζεστε την γεωργία στην Ευρώπη αναφέρεται στις συνθήκες ότι η επιστηστική ασφάλεια πρέπει ε, να είναι μέλημά μας. Και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην περαιτέρω διαμόρφωση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το περιβάλλον και η γεωργία πρέπει να συνδυάζονται, αλλά ε, πρέπει να είναι σαφές ότι και η κοινωνική πολιτική παίζει ρόλο στην Ήπεθρο, γιατί αυτό σημαίνει για μένα, στη τελευταία ανάλυση, ότι έτσι μόνο μπορούμε να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα. Θέλουμε όλοι να εργαστούμε περισσότερο για αυτά τα τρία θέματα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η χρηματοδότηση, η διοίκηση και ο έλεγχος θα είναι θέματα για τα οποία θα είμαι ε, εισηγήτρια, αλλά στο Συμβούλιο έχει κολλήσει η κατάσταση. Και δεν είναι σαφής και ο προϋπολογισμός που θα έχουμε. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, απευθείας η ερώτησή μου σε εσάς, Πότε θα υπάρξει αυτός ο μεταβατικός κανονισμός. Χρειαζόμαστε αυτό το, το μεταβατικό κανόνα. Πότε θα υποβάλλετε την πρόταση αυτή και για ποιο χρονικό διάστημα θα ισχύσει. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ρωστούμε παράλληλα. Γιατί όποιος είναι ρεαλιστής διαπιστώνει ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται πριν το 23. Άρα πρέπει να μπορούν να προγραμματίσουν ε, τη δουλειά τους οι, οι γεωργοί. Χρειάζεται ένας νέος ε, μεταβατικός κανόνας για να περάσουμε από τη συμμόρφωση προς την απόδοση. Και μας ανησυχούν και μεταφορές ε, ζών των ζώων προς τα σφαγεία. Και το Μερκοσούρ, 99.000 ε, τόνοι, ναι 1% αλλά άμα δείτε τώρα τα τμήματα, κοιτάξτε τα τμήματα των ζώων δηλαδή, είναι τα πιο πολύτιμα και η αξία τους είναι 15%. Παρ' όλα αυτά, οι γεωργοί στη χώρα μου ανησυχούν ιδιαίτερα για το πώς διεξήχθη ο δημόσιος διάλογος. Και φυσικά και για την προκλήση, τις προκλήσεις που προκύπτουν από το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χόισλινγκ. Καλό που είστε εδώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι πρέπει να μας υποβάλλετε ένα κείμενο για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Υπάρχει η έκθεση για την τρομερή μείωση της ε, βιοπικιλότητας, όπου συμβάλλει και η Γεωργία. Έχουμε επίσης ε, ένταση της κλιματικής αλλαγής. Και το σχέδιό σας, στην ουσία τι μας λέει, όπως και πριν τα πράγματα, κυρίως πληρώνουμε με βάση τις επιφάνειες. Και όχι βέβαια σε όλους, αλλά κυρίως στους μεγάλους γεωργούς. Ε, δεν είναι αυτή η πολιτική ε, προσαρμοσμένη στην κατάσταση. Πραγματικά ίσως θα έπρεπε να αποσύρετε και να την ξαναρχίσετε από την αρχή αυτή την πρόταση. Και τώρα, επιπλέον, συμφωνία Μερκοσούρ. Πριν από τρει μήνε είπατε, καλά δεν θα είναι τόσο άσχημα, αλλά είναι χειρότερα από ό,τι φοβόμασταν. Έχουμε και τι ποσοστό για τα πουλερικά μα λέτε δεν είναι και τόσο πολύ, 99.000 ε, βόλιο. Ναι, αλλά με τον Καναδά είχαμε 50.000, με τι ΗΠΑ έχουμε 30.000 τόνου. Αυτά σε μερικά χρόνια θα καταστρέψουν την αγορά βοήθεια. Τα ξέρετε και από τη χώρα σα, όπου ε, σα επικρίνουν πολύ έντονα. Και λέτε, ναι, θα φροντίσουμε να τηρηθούν και οι συμφωνίε των Παρισίων για το κλίμα. Μα μας λέτε ότι δεν υπάρχει παράνομη αποψήλωση των δασών στην ε, Βραζιλία. Μα είναι αστεία αυτά. Δεν είδατε τα νούμερα. Είδατε ότι η παράνομη αποψήλωση τώρα νομιμοποιείται από τον Μπολσονάρο. Το είπε προχτές. Οι Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να αναμειχθούν από την δική μας εσωτερική πολιτική. Με αυτόν κάνετε συμφωνίες. Είναι σκανδαλώδες. Κοιτάξτε. Μας λέτε ότι είναι τόσο θετικά όλα αυτά. Είπατε ότι θα τους εξάγουμε περισσότερες σοκολάτες. Θα ευχαριστηθούν οι Ευρωπαίοι Γεωργοί γι' αυτό. Είμαστε θύματα μιας πολιτικής που θέλει να πουλάει πρώτα απ' όλα βιομηχανικά προϊόντα. Και η Γεωργία ξεπουλιέται γι' αυτό. Λέτε ότι είναι καλή αυτή η συμφωνία. Γιατί θα πληρώσετε δισεκατομμύρια για αποζημιώσαμε τόσο καλή αυτή η συμφωνία. Για εξηγήστε μας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ντάβιντ. Από ό,τι άκουσα μπορώ να μιλήσω τσεχικά, επομένως ε, θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική έχει αυξήσει τις ανισότητες και έχει οδηγήσει σε πτώση της παραγωγής. Η ανάπτυξη της υπαίθρου και η γεωργία έχουν φτάσει σε αδίέξοδο. Τα γεωργικά αγαθά είναι στρατηγικής αξίας για κάποιες χώρες. Έχουν σχέση και με εθνική ασφάλεια και ε, κοινωνική ανάπτυξη στην Ήπεθρο. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Λετωνία έχω δει χωριά τα οποία ε, ε, ξοντώθηκαν καθαρά, ξεκάθαρα και δεν υπάρχει καμία καλλιέργεια στη γη και ε, δεν έχουν μετατραπεί σε βοσκοτόπους ή σε δάση. Απλώς είναι καλυμμένα ε, με ζυζάνια. Σε 30 χρόνια στην Τσεχική Δημοκρατία είδαμε πτώση στην απασχόληση στον τομέα της γεωργίας εν μέρη λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά κυρίως λόγω της κατάρρευσης ε, της ε, ε, κτηνοτροφίας. Υποβάθμιση του εδάφους και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία ορισμένες φορές. Υπάρχει μια άνηση προσέγγιση στην οικονομία της υπαίθρου. Η εμπορική συμφωνία με το Μερκοσόρ απλώς θα επιδεινώσει τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Δεν πρόκειται για ευκαιρία, αλλά για απειλή. Βλέπουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και γι' αυτό ακριβώς ε, σκοπεύουμε να είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί και δεν θα δεχτούμε αλλαγές οι οποίες θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Δεν έχω καμία ερώτηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Α, η κυρία Μάκινταρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ σήμερα. Είμαι στο πίσω μέρος της αίθουσας πλέον. Απόλαυσα τη συνεργασία μας σε όλη την προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι έχουμε πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Τα αναφέρατε κάποια εξ αυτών, αλλά εγώ επειδή πάντα είμαι υπέρμαχο των μικρών γεωργών και των μικρών επιχειρήσεων, είμαι ιδιαίτερα περήφανη για την οδηγία για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Θεωρώ ότι πρόκειται για τεράστιο άλμα και μάλιστα οι περισσότεροι γεωργοί είναι μικρές επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι μειώσαμε το διοικητικό άχθος για αυτούς ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτική σημασία. Τα περιθώρια στη γεωργία είναι πολύ μικρά και επιπλέον κόστος πραγματικά απειλεί την επιβίωση κάποιων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων η τεχνολογική πρόοδος στη γεωργία μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικότερη και βιωσιμότερη γεωργία και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να βρισκόμαστε στην αιχμή της ε, γεωργικής τεχνολογίας, σε καινοτομίες και σε σταθερότητα. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε ότι ε, τα ωφέλη της τεχνολογικής καινοτομίας θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους γεωργούς, μεγάλες, μικρά, ε, όσοι κάνουν συμβατική γεωργία, βιολογική γεωργία, οι τεχνολογικές λύσεις ε, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και για τους μικρούς γεωργούς αλλά και για τους μεγαλοκτηματίες. Επομένως, ε, η ερώτησή μου είναι πώς βλέπετε ότι θα υπάρξει πρόοδος στην τεχνολογία της γεωργίας για βιώσιμη γεωργία. Πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο σε αυτά στο διάρκεια της επόμενης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Δυστυχώ η πρόβλεψή σα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα παίζω γκολφ ε, μετά τι ευρωεκλογέ ε, δεν παληθεύτηκε και είμαι βέβαιο ότι είστε σίγουρο, χαίρεστε που είμαι εδώ σήμερα. Εγώ και ο συνάδελφος ρωτήσαμε την ε, Επιτροπή για το Βόηο Κρέας ε, ε, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και μου είπατε για ό,τι θέλετε αρκεί να μην είναι αποζημίωση για το Brexit. 50 εκατομμύρια ευρώ των φορολογουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείωση της παραγωγής ήταν μία από τις επιλογές οι οποίες ήταν διαθέσιμες. Η μείωση της παραγωγής είναι αυτό το οποίο επέλεξε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Η μείωση του βόηου κρέατος που παράγεται σε μόνιμους βασκοτόπους με υψηλά πρότυπα ευημερία των ζώων, δηλαδή πρόκειται για βόλιο κρέα ε, ε γάλακτο. Ε, Επομένω, ε, μετά από αυτό έρχεται και η συμφωνία του Μερκοσούρ για 99.000 τόνου εισαγόμενου που θα είναι οτιδήποτε εκτό από βιώσιμο βόλιο κρέα. Σήμερα εξελέγει ο Μπόρι Τζόνσον ως ε, πρόεδρος των συντηρητικών και κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη θα γίνει πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ξέρετε κύριε Επίτροπε, η Ιρλανδία ε, εξάγει 250.000 τόνους ε, το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν προχωρήσουμε τον Brexit, τότε οι Ιρλανδοί αγρότες, και κτηνοτρόφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αρμαγεδόνα. θα χάσουν πρόσβαση στην πιο σημαντική του αγορά σε μια χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται γιατί δίνεται δίνετε χρήματα στην Ιρλανδία, επομένω το δέχεστε, ότι πιέζονται οι κτηνοτρόφοι βόλου κρέατο. Πώ είναι λογικό λοιπόν να εξετάσετε μια τέτοια συμφωνία. Όπω μου είπε ένα κτηνοτρόφο, εξηγήστε γιατί ε, προσφέρετε μια ασφάλεια 50 ε, εκατομμύρια ευρώ τη μία εβδομάδα στην Ιρλανδία και τώρα την επόμενη εβδομάδα του το κόψατε και κατά πάσα πιθανότητα ε, θα καταρρεύσει. Πραγματικά εξηγήστε μου γιατί γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Οπότε κλείσαμε τους συντονιστές. Οπότε ο κύριος Επίτροπος για να απαντήσει. Θα πρότεινα ε, ιδανικά κύριε Επίτροπε πέντε λεπτά. Γιατί είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι υπεραιτέρω που θέλουν να ρωτήσουν. Αλλά βλέπετε κύριοι συνάδελφοι, το λέω για τους νέους, είναι πολύ ζωαρή, ζωηρή συνόμη συζήτηση. Νομίζω ότι έχει πολλά να μας πει ο κύριος ε, Επίτροπος, ε, κρίνοντας και από, αυτά που μας, ε, από τις εκφράσεις του προσώπου του. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά τους συντονιστές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Θα ήθελα να συνδέσω τα σχόλια που κάνετε για το οικονομικό σκέλος, τα χρήματα και τις πολιτικές. Α, όπως είπατε πολλοί από σας. Όλοι θα θέλαμε βεβαιότητα και για τους αγρότες μας και για τους πάντες. Αν καταλήξουμε σε συμφωνία για το οικονομικό σκέλος ε, και ολοκληρώσουμε και διεκπαιρεώσουμε τις συνομιλίες για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στο τέλειο έτος. Αλλά φαντάζομαι ότι όπως και στο παρελθόν θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ε, και αν υπάρχει πολιτική βούληση θα μπορέσουμε να έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Και το ίδιο θα κάναμε αν είχαμε ιδέα ήδη για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και το γεωργικό προπολογισμό, τον προπολογισμό τη ΚΑΠ. Οπότε η ιδέα ενό μεταβατικού κανονισμού ε, δεν μα βρίσκει ξένου. Είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που χρειαστεί, αλλά προτιμούμε να διεκπαιρεώσουμε τα θέματα αυτά το φθινόπωρο στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να προοδεύσουμε όσο γίνεται και το φθινόπωρο θα κάνουμε νέα αξιολόγηση. Θέλουμε όμως να ε, διαβεβαιώσουμε τους αγρότες μας, κάτι που θέλετε κι εσείς, ότι θα συνεχίσει η ροή των κονδύλιων προς τους αγρότες, άσχετα με το χρονοδιάγραμμα των συμφωνιών και των α, ρυθμίσεων. Το θέμα του γεωργικού ισοδύναματος είναι ύψητη προτεραιότητα. Δεν θα πρέπει να είναι υποδέστερο σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες και τα διαδικαστικά ε, στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κύριε Χόισλινγκ, φαντάζομαι θα σα εκπλήσει το γεγονό ότι δεν έχω καμία πρόθεση να αποσύρω τη συμφωνία. Πάντω, σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε για τη συμφωνία, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και αποδεχόμαστε ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξία στο κλίμα και το περιβάλλον. Και μάλιστα ήταν διπλάσιε οι φιλοδοξίε που είχαμε με βάση την τελευταία πρόταση για το περιβάλλον και το κλίμα. Θα πρέπει όμως να δούμε τα πράγματα σε αυτό το νέο πλαίσιο και τις νέες απαιτήσει ε, που έχει η κοινωνία μας από όλους τους τομείς που θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους και για τη κτηριακή πολιτική, για την απόδοση των κτηρίων, τη γεωργία, τις μεταφορές. Θα πρέπει όλοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των στόχων, όχι απλώς να τα λέμε στη θεωρία, όπως πολλές φορές έγινε στο παρελθόν. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να υλοποιούμε τους στόχους. Και Περιμένω τις προτάσεις σας παλιούς από παλιούς και νέους ευρωβουλευτές για να έχουμε προγράμματα ρεαλιστικά και πρακτικά για να μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς μας στόχους με τη συμβόλη και της γεωργίας. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι η έννοια, η ιδέα ότι ε, το, η συμφωνία του Μερκοσούρ θα είναι θετική για τη Γεωργία, ε, όντως ε, είναι κάποια, κάπως προβληματική. Αυτό το ξέραμε από την αρχή. Αλλά με βάση την εντολή που λάβαμε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε πολύ αμυντικοί στη Γεωργία. Όπω σα είπα, με τι συμφωνίε που κάναμε για το Βόιο, το πουλερικά και άλλου κλάδου στη ζάχαρη, για μερικού τομεί, όπω ε, τα ενοπνευματώδη, τα μπελονικό τομέα, προστασία των γεωρικών ε, ε, ενδείξεων. Ήμασταν πολύ πιο προστατευτικοί, αλλά σε μερικά θέματα, σε μερικού τομεί είχαμε απελευθέρωση, όχι πλήρη σε όλου. Και είχαμε πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε. Προσπαθήσαμε να μετριάσουμε αφενό τι ποσότητε και αφετέρου να ε, επεκτείνουμε τη μεταβατική περίοδο, να την παρατείνουμε ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, δεν μας είπατε τίποτα για τη θετική έκβαση των συμφωνιών με την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Εκεί πραγματικά αντισταθμίσαμε την εισαγωγή προϊόντων μέχρι 65.000 ε, ε, τόνους από την Ιαπωνία, 40.000 ε, τόνους προϊόντων από το Μεξικό και εκεί θα ολοκληρώσουμε τις νομικές πτυχές του χρόνου, όλες αυτές οι εξελίξεις ήταν θετικέ για τους αγρότες. Και ανοίξαμε την ε, αγορά της Κίνας που ήταν πολύ δύσκολη για πολιτικούς λόγους και όχι για λόγους ασφάλειας τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μερικές ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν επιτυχώς να έχουν πρόσβαση στην κινέζικη αγορά. Και τώρα ε, η Κίνα δεν ε, αντιμετωπίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο εταίρο για την εμπορία επιλεκτικά ανοίγει τι αγορέ τη σε συγκεκριμένες χώρες όπως τη Γαλλία και τις Κατοχώρε. αλλά 10.000 τόνοι το χρόνο είναι το έλλειμμά τους από πρωτενε. και αυτή τη στιγμή από, κυρίως ε, φοδιάζονται από την Νότια Αμερική για τις πρωτεΐνες ενώ εμείς με τα υψηλά Υψηλή ποιότητα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το έλλειμμα που έχει η Κίνα. Σε ό,τι αφορά την ισορροπία τη αγορά βοήου κρέατος, έχουμε 105.000 τόνου που θα τύχουν άμεση εφαρμογή στην τελε... επόμενη διετία, όταν θα έχουμε χρόνο να προσαρμοστούμε στους 99.000 επιπλέον τόνους ε, που ε, θα εισαχθούν αν δεχθεί αν δεχθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την συμφωνία αυτή του Μερκοσούρ. Και αυτό θα γίνει σε έξι ετήσιες φάσεις, όπως σας είπα. Ε, και αυτή τη στιγμή 270.000 τόνοι ε, που είχαμε από προηγούμενες συμφωνίες ε, τη χάνουν επιτήρηση επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχου. Και πολλές χώρες όπως η Ιρλανδία, όπου το 2018 δεν είχαμε κανένα προϊόν βοηοκρέατος που δεν πήγε απευθείας στην Ιρλανδία. Το 2018 δεν είχαμε καμία τέτοια άμεση εισαγωγή από τις χώρες του Μερκοσούρ. Οπότε θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά με βάση τα πραγματικά περιστατικά, τα γεγονότα. Και σίγουρα η συμφωνία, αν είχε τόσο αρνητικά αποτελέσματα για τη Γεωργία όπως αυτά που λέτε μερικοί, θα την υπέγραφα. Και για πρώτη φορά, όπω σα είπα, έχουμε κονδύλιο ενό δισεκατομμυρίου για την υποστήριξη τη γεωργία. Σε περίπτωση που υπάρχει στρέβλωση ή διαταραχή τη αγορά, μπορεί να το αποφύγουμε. Αλλά για πρώτη φορά έχουμε προβλέψει ειδική χρηματοοικονομική υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο κλάδο, για τη γεωργία. Και ένα μηχανισμό με ασφαλιστικέ δικλείδε που αρχικά είχε προταθεί από την Γαλλία για τα TRQs, για τι δασμολογικέ ποσοστώσει μέχρι στιγμή δεν υπήρχαν. Και Νομίζω ότι τηρήσαμε τις προδιαγραφές και τα υψηλά μας πρότυπα. Κύριε Φλάναγκαν, δυόμιση ώρες αφιερώσαν πάλι μου στη γενική μας διεύθυνση για να σας εξηγήσει ε, ποια είναι τα θετικά για την Ελλανδία του Βορείου Πακίτου. ε, αν πραγματικά κάτι τέτοιο επιθυμούν η εκλογή σας, η γεωργή σας, πείτε το. Αλλά νομίζω ότι τα παρα, παραπλανητικά μας τα πα, παρουσιάσατε. Και αν είναι πραγματικά κάτι τέτοιο αυτό που θα επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Αλλά θυμάμαι παλιά πως ήταν πολύ πιο ισχυρός υπέρ του περιβάλλοντος υπέρμαχος. Ευχαριστώ. 34 συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ζητήσει το λόγο. 34. Μπορώ να κλείσω το κατάλογο. Υπάρχει κανένα άλλο. Ωραία, κλείνει ο κατάλογο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα. Και τονίζω. Ένα λεπτό. Πρώτο. Ο συνάδελφο Κάζη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Εγώ ποτέ δεν υποτίμησα τις δυνατικέ σα ικανότητες και την πονηριά σα. Το 2016 μάλιστα σε, στις ε, εφημερίδες λέγατε ότι το βόλιο κρέας δεν θα ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με Μερκοσούρ. Είχα πει τότε στις ε, γεωργικές οργανώσεις ότι τους κοροϊδεύατε για να μην αντισταθούν στη συμφωνία θεωρώντας ότι το βόλιο δεν θα συμπεριληφθεί και τελευταία στιγμή θα τους τη φέρετε. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Οι γεωργοί δεν θέλουν ε, αποζημιώσεις. Θέλουν να κερδίζουν χρήματα από τα προϊόντα τους, που είναι το καλύτερο βόλιο στον κόσμο το δικό μας και τα καλύτερα πουλερικά. Οπότε, κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μπουρδες για την ε, αποδάσωση που λέτε στις χώρες Μερκοσούρ. Τι περιβαλλοντική έννοια έχει να μεταφέρεις 100.000 τόνους βόλου από την άλλη άκρη του κόσμου για να αντικαταστήσεις το πιο βιώσιμο και υψηλότερη ποιότητα βόλου που παράγουμε εμεί εδώ στην Ευρώπη. Μπορείτε παρακαλώ να απαντήσετε αυτή την απλή ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω. Ένα λεπτό παρακαλώ. γιατί αλλιώς θα πάρουμε πολύ χρόνο. Η κυρία Αβραάμ. Χαίρετε κύριε Επίτροπε, Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την παρουσίασή σας. Δυστυχώς ε, και εγώ πρέπει να εκφράσω τις ανησυχίες μας, ε, όπως και, τις ανησυχίες μου, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, για τις αρνητικές επιπτώσεις της Συμφωνίας Μερκοσούρ για τη Γεωργία διαφόρων χωρών της Ένωσης και της Ρουμανίας, αλλά και για τη δική σας χώρα. Γιατί μετά από δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει ενημερωμένη μελέτη αντικτύπου. Έχουμε βέβαια αυτό το δίκτυο ασφαλείας ενό δις ευρώ. Είπατε λοιπόν ότι μπορεί να πάνε λάθο τα πράγματα, μπορεί να πάνε στραβά τα πράγματα. Γιατί όμως, γιατί όμως ε, ζητάτε αυτή τη χρηματοδότηση και από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Και δεύτερον, πώς μπορείτε με συγκεκριμένα στοιχεία να καθησυχάσετε του γεωργού μα ότι θα επιζήσουν γιατί τους έρχονται τα προϊόντα του Μερκοσούρ. Ε, γίνονται περικοπές του προπολογισμού και επίσης υπάρχουν και άλλες προτιμησιακές συμφωνίες, σε άλλες ε, ε συμφωνίες ελευθερών Υπάρχει και κλιματολογική απειλή και έχουμε και τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και βιώσιμη γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντριού. Χαίρομαι που βλέπετε, βλέπω ότι είστε σε φόρμα κύριε Επιτροπέ, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι μήνυμα και στείλουν εκλογή εσείς είστε σταθερός. Παρά τον Brexit, παρά τη ΣΕΤΑ, 100.000 σε Έχουμε τη συνεχή μείωση των προπολογισμών. Έχουμε τα ελλείμματα για τις πρωτεΐνες και για τα φυτικά προϊόντα. Και κοιτάξτε για το Μερκοσούρ. Σας παρακαλώ να μην κάνετε επίσημα ταξίδια να πάτε στι χώρες που είναι η ουσία του προβλήματος. Πήγαμε ω αντιπροσωπεία στο Μάτο Γκρόσο. Και αυτό που είδαμε πραγματικά δεν είναι αυτό που μας περιγράφεται. Και τα σκάνδαλα που είδαμε στη Βραζιλία δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζεται. Εγώ θεωρώ ότι οι ρήτρε διαφύλαξης που προβλήπονται στη συμφωνία είναι σαφώ ανεπαρκείς. Και το λέτε και εσεί. Προβλέπετε ένα δι που θα μπορούσε να αποδεσμευθεί εάν υπάρξουν αναταραχές στις αγορές. Μα πώς δυνατόν να κάνετε και τον πυρομανή και τον πυροσβέστη. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής που έχουμε υποχρέωση να ε, προστατεύσουμε συλλογικά. Ευχαριστώ πολύ. Σφάια Πύρικ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας. Πρέπει φυσικά να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι ήρθατε ε, και μας εξηγήσατε ε, τελικά την κατάσταση και αυτό δεν μας κάνει αισιόδοξου και το βόλιο και το χείριο κρέας. Πώς είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι πάνε καλά. Αυξήθηκαν οι ποσοστώσεις από 80 στα 180.000 τόνους για τα πουλερικά και για τα κατανοητικά προϊόντα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που αφορούν το σύνολο των τομέων. Είπατε ότι υπάρχουν κάποια ποσά διαθέσιμα. Αλλά το ΚΟΠΑ, ΚΟΖΕΚΑ και οι διάφοροι οικονομολόγοι μας λένε ότι μπορεί να φαλήρουν 2.000 επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια. Και άλλη μια ερώτηση. Ελπίζω να απαντήσετε. Τι αναμένετε από το διάλογο με τους υπέρμαχους της ευημερίας των ζώων στις χώρες Μαρκοσούρ. Ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ζέστη στις Βρυξέλλες. Θα γίνει 35 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο και 38 βαθμούς στο λιμάνι της Τζέντα. Και εκεί έχουμε ένα σκάφος με 17.000 πρόβατα έφυγε από τη Ρουμανία και πηγαίνει στο Κουβέιτ αυτό το καράβι και πρώτη φορά ένα τέτοιο μεγάλο σκάφος ε, να χωρεί από την Ευρώπη και ε, έχει κατεύθυνση τον Περσικό κόλπο. Τα ζώα θα πεθάνουν επί του σκάφους και θα πεθάνουν στο Κουβέιτ γιατί ε, εκεί δεν έχει 38 βαθμούς, έχει 48 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες έγιναν κάποιες απόπειρες να μην ε, αναχωρήσει, αλλά συνεχίζει την πορεία του. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ο Επίτροπος Ανδρουκάουτες ε, είπε ότι αυτή είναι πολύ βάναυση μεταφορά ζώων. Αυτό λοιπόν ε, κρύβεται πίσω από αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Θα κάνετε κάτι για να υπάρξουν διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ρουμανίας. Κύριε Αγγιλέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Χόγκαν, καλωσορίσατε. Μα ανησυχεί το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ο προπολογισμό. Δεν ξέρουμε πώς ε, θα ε, οριστικοποιηθεί τελικά. Οι περικοπές για την ανάπτυξη της υπαίθρου δεν μας αρέσουν και σε μένα προσωπικά και νομίζω ότι και στην ομάδα μου ε, είναι καλύτερη λύση, θεωρούμε ότι είναι καλύτερη λύση η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιστοίχω και για τον Brexit. Η κατάσταση δεν βοηθά καθόλου και με τον Μπόρις Τζόνσον που ανέλαβε τα Ινία ε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι καλύτερο. Όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, ε, μας, ανησυχεί κυρίως, μας ανησυχεί κυρίως το Μερκοσούρ, αλλά το θέμα είναι ότι η αρχή της ισοδυναμίας ίσως να μην αρκεί για τις συμφωνίες ε, και την αμοιβαιότητα. Διότι βλέπουμε ότι τα διάφορα μοντέλα παραγωγής έχουν μεγάλο αντίκτυπο για κάθε κλάδο. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει ανησυχία. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να μου πείτε ε, τι θα γίνει με τις τιμές ε, του ελαιολάδου στην Ισπανία που μειώνονται. Θα ληφθούν κάποια τα μέτρα που πρότεινε η χώρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νόχελ. Ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας. Στην ε, ομιλία σας άκουσα ότι εσείς πρέπει να ήσασταν επίτροπος εμπορίου. Εσείς δεν μιλάτε για γεωργία, μιλάτε μόνο για εμπόριο. Η γεωργική πολιτική δεν είναι μόνο εμπορική πολιτική. Και κάτι άλλο. Ξεχάσατε να ακούσετε Συγγνώμη, ξεχάσατε να δώσετε σε ένα σημείο μα στην κυρία Φόντερ Λάιεν, γιατί στην ομιλία τη δεν είπε ούτε κουβέντα για τη Γεωργία. Δεν είναι δυνατόν κάποιο να εκλέγεται πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί να λέει τίποτα για τη Ουρία. Δεν ξέρω. Οι άλλοι επίτροποι τη δώσαν τι να πει, εσεί δεν τη είπατε. Δεν τη δώσατε τίποτα. Θα ήθελα να μα πείτε τι θα κάνει για τη Γεωργία κυρία Φόντερ Λάιεν. Τώρα για το Μερκοσούρ. Πολύ περίεργο είναι να αντιμετωπίζετε αρνητικά η συμφωνία για το Μερκοζούρ από τους Γιώργους. Ενώ άλλες συμφωνίες ε, για τη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, αντιμετωπίζονται θετικά, παρά το ότι οι γεωργοί έχουν άλλη άποψη. Και απέναντι είναι πολύ λυπηρό ότι στηρίζεται αυτή τη συμφωνία Μερκοσούρ. Ο Σάλφος ο Λέκας. Ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Εγώ είμαι νέο μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, οπότε δεν θα είμαι τόσο επικριτικός όσο κάποιοι προλαλήσατε συνάδελφοι. Φαίνεται εκείνοι σας τα έχουν μαζεμένα από προηγούμενες θητείες. Συμφωνώ πάντως ότι ο γεωργικός κλάδος θα πρέπει να είναι βιώσιμος, να εστερνιστεί την τεχνολογία, την έρευνα και την ε, καινοτομία και τα προϊόντα, τα γεωρικά προϊόντα να είναι υγιεινά και υψηλής ποιότητας. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε και θεμητό ανταγωνισμό. Είναι γνωστό ότι θεμητός ανταγωνισμός δεν υπάρχει ούτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, άμεσες ενισχύσεις. Το γνωρίζετε. Οι γεωργοί της Βαλτικής και κυρίως οι Λιθουανοί αγρότες έχουν πολύ χαμηλότερες κρατικές ενισχύσεις από ότι γεωργοί άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε πώς μιλάμε για δίκαιο ανταγωνισμό, για θεμητό ανταγωνισμό. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στις δημοσιονομικές προοπτικές. Στο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει ε, στα πλαίσια των οικονομικών ρυθμίσεων να επιλύσουμε και το θέμα της αδικίας που ισχύουν μεταξύ των Ευρωπαίων Γεωργών για τις άμεσες ενισχύσεις. Κυρία Κατάινεν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την ε, παρουσίαση που μας κάνατε. Για το Μερκοσούρ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε ένα δισεκατομμύριο για τους ε, γεωργούς που θα ε, υποστούν ζημία από τις εισαγωγές από τις χώρες του Μερκοσούρ από πού θα βρεθεί αυτό το 1 δισεκατομμύριο, από τους μηχανισμούς διαχείρισης των κρίσεων ή θα είναι ένα ξεχωριστό κονδύλιο. Και επίσης, ε, γιατί προβλέψατε αυτή την επιχορήγηση, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχω καταλάβει. Θα πρέπει να προβλέψουμε φυσικά ε, συμπληρωματική ενίσχυση για τους γεωργούς, γιατί θα είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός που θα υποστούν από τις χώρες του Μερκοσούρ. Για τη Ρωσία είχαμε σχετικά άμεση επιβολή των ε, κυρώσεων. Το Μερκοσούρ όμως είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία η σχετική εμπορική συμφωνία. Επίσης, ποια θα είναι η μεταβατική περίοδος για τη μεταρρύθμιση ΚΑΠ, ένας χρόνος ή μήπω μια διετία. Ευχαριστώ κύριο Σαβαρμά. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω κύριε Επίτροπε εδώ, ακμεότατο όπως πάντα. Την προηγούμενη πενταετία ασχολήθηκα με τον προϋπολογισμό και γι' αυτό θα σταθώ στο δημοσιονομικό σκέλος και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει πίεση για περικοπές, ειδικά στο γεωργικό προϋπολογισμό. Με ενδιαφέρει όμως η δική σας άποψη για το σχόλιο μου. Σίγουρα υπάρχουν πολλά εύλογα επιχειρήματα ε, ε, υπέρ τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση για την κοινή γεωργική πολιτική. Και πρώτο βασικό επιχείρημα είναι το περιβάλλον, το κλίμα μάλλον. Αν θέλουμε όντω σοβαρά να βάλουμε τη γεωργία μα και του αγρότε μα στην πρώτη γραμμή του πολέμου για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να του εξασφαλίσουμε τα μέσα και του πόρου για να το κάνουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από του γεωργού ταυτόχρονα να παράγουν ε, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και ταυτόχρονα να είναι και στην πρωτοκαθεδρία ε, στα κλιματικά ζητήματα. Δεν μπορούν ταυτόχρονα να παίζουν σε όλα τα ταμπλό οι Γεωργοί μας χωρίς υποστήριξη. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Ξέρω ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως στο Μερκοσούρ και μας προβληματίζει για το μέλλον. Τι γίνεται όμως με την παρούσα κρίση που αντιμετωπίζει το μέρο του βοηού κρέατο, που είναι και πραγματική και άμεση. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη πτώση τη τιμή του βοηού κρέατο, υπάρχει πρόβλημα στην κατανάλωση και από ό,τι φαίνεται και στην, στον ανεφοδιασμό, στην προμήθεια. Γιατί ε, μιλήσετε για μία δεκαετία, αλλά η κρίση είναι εδώ και τώρα για του γεωργού. Οπότε υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης στο Βόλιο και αν ναι, τι πρωτοβουλίες περιλαμβάνει. Ευχαριστώ κύριο Σαμάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να σταθούμε και στο εξή θέμα. θα θάτερον, όπως λέμε και στην Πορτογαλία. Ή η γεωργία θα θεωρηθεί στρατηγικό τομέα ή όχι. Και αν δεν είναι, το, αν είναι στρατηγικό τομέα, δεν επιτρέπονται περικοπέ ούτε στι ενισχύσει, ούτε στην αγροτική ανάπτυξη. Υπάρχει και το θέμα τη κυριαρχία των κρατών μελών. Της, γιατί μιλούμε για παραγωγή, για παραγωγή τροφίμων και για ασφάλεια τροφίμων. Ε, και επειδή έχουν και νέες προκλήσεις οι γεωργοί να αναλάβουν περιβάλλον και κλίμα, θα ήταν απολύτω άδικο να έχουμε περικοπές στη γεωργία. Σε ό,τι αφορά το Μερκοσούρ, ε, μιλήσετε για ένα δισεκατομμύριο βοήθεια για, σε περίπτωση διαταραχής της αγορά. Αυτό όμως είναι πολύ γενικό και όριστο. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη θέση και κατάστη, ε, άποψη της κατάστασης αναχώρα και αναγεωργία, ανατομέα. Έτσι θα μπορούμε να λάβουμε θέση για τη συμφωνία αυτή. Κυρία Σαντέρ, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω στο ζήτημα του Μερκοσούρ και να σας εκφράσω την ανησυχία μου και την προσωπική αλλά και των Γάλλων και Ευρωπαίων Γεωργών. Κύριε Επίτροπε, πώς θα καθυσυχάσουμε τους Γεωργούς μας, πώς ε, θα μεριμνήσουμε για τις ανησυχίες, να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες των τευτελοπαραγωγών, των ε, βοοτρόφων και των ε, πτηνοτρόφων μας. Πώς θα τους καθησυχάσουμε. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα. Ασφαλιστική δικλίδα σε περίπτωση αποσταθεροποίησης αγορά. Πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι θα ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα αμέσω, γιατί έχουμε και το παράδειγμα του ρυζιού πρόσφατα. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα εφαρμόσετε αυτό το ε, σχέδιο στήριξη ενό δισεκατομμυρίου και σε ό,τι αφορά την υγειονομική κατάσταση και την ε, αξιοπιστία των ε, ελέγχων στι χώρες του Μερκοσούρ. Εξακολουθεί να είναι ενισχυτική κατάσταση για τους υγειονομικούς ελέγχους. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε και να μας καθησυχάσετε. Πάντω για τη συμφωνία αυτή με το Μερκοσούρ, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην προτείνετε μεταβατική της εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μόκλερ. Ευχαριστώ. Εγώ συμμερίζομαι τις ε, επιφυλάξεις για το Μερκοσούρ και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος και πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά δεν απαιτούμε από τους εταίρους μας ε, παρόμοιες ε, εγγυήσεις ε, σε εμπορικές συμφωνίες. Είναι σωστό αυτό. Εντάξει, είπαμε ότι το Brexit θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο για τους Ιρλανδούς, αλλά για όλους τους γεωργούς και εκτενοτρόφους της Ένωσης. Και έχουμε το γεγονός ότι για τους γεωργούς μας υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Η κοινή γεωργική πολιτική ήταν πάντα βασικός ε, κινητήρας της ε, ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το βασικό θέμα, επιστηστική ασφάλεια, να μην υπάρχει πείνα, να μην τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Να τα λαμβάνουμε υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Πρώτη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις συνέπειες της ξηρασίας για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Σε τι βοήθεια μπορεί να βασίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από την ξηρασία. Στη συνέχεια, Μερκοσούρ. Πρόκειται για εμπορικέ συναλλαγές οι οποίε αξίζουν ε, δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά οι γεωργοί μα θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο, ε, κυρίως κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με βόηο, κρέα πουλερικά ε, ή και την εθανόλη. Στην Πολωνία οι γεωργοί αναφέρουν 20% μείωση στι τιμέ. Μειώθηκε η περιοχή ε, ε, ε, για την βιοθανόλη. Ελπίζω να αλλάξει το θέμα σύντομα. Ο Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ανησυχώ για το μέλλον τη συμφωνία Μερκοσούρ. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι επιζήμια για του γεωργού μα. Κύριε Επίτροπε, στην αρχή προσπαθήσατε να είσαστε καθησυχαστικό και μετά μα είπε ότι υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλεία ενό δι ευρώ, που σημαίνει ότι συνειδητοποιείτε του κινδύνου, ιδίω για την παραγωγή βόλου ε, κρέατο και τελικά παραδεχτήκατε ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε σε όλου του τομεί. Και εν τέλει, εδώ συνοψίζω αυτά που μα είπατε και θα ήθελα απλώ να το επιβεβαιώσω. Μα λέτε ότι με τη συμφωνία για το Μερκοσούρ μειάσατε το βόλιο κρέα ε, προ όφελο των εξαγωγών για τα ενοπνευματώδη ποτέ. Και αυτό πρέπει να σα πω ότι με σοκάρει. Έχω και μία πιο συγκεκριμένη ερώτηση για την ξηρασία σε μεγάλο τμήμα τη Γαλλία, η οποία πλήττεται αυτή τη στιγμή. Ο Υπουργό Γεωργία σα ζήτησε να δώσετε προκαταβολή από 50% έω 75% που θα δοθούν τα μέσα Οκτωβρίου. Θα ήθελα να ξέρω αν είστε διατεθειμένο να δεχτείτε αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ κυρία Πυρμπάκας. Έκτος μικροφώνου κυρία Πυρμπάκας. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας συναντώ ως ε, νέα Ευρωβουλευτής από τις υπερπόντιες ε, περιοχές. Να σας πω ότι καταρχώς ε, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, έχουμε και τη Ριουνιόν και τη Μαγιότ για τα τρει υποπτέ περιοχές έχουμε τη Μαρτινίκα, τη Γουαδελούπη, το, ε, τη Ρεουνιόν και ξέρετε τι γίνεται με τη χρηματοδότησή τους ε, για τη Γουαδελούπη, για τη Μαρτινίκα, για τη Σύμβαση των Κανών που πηγαίνει μέχρι το 2022. Μετά το 2022 τι θα υπογίνουμε εμείς οι γεωργοί της Γουαδελούπης, ε, της Ρεωνιών και της Μαρτινίκας για να μπορέσουμε να επιβεώσετε Ξέρετε ότι εμείς ζούμε από τη γεωργία, από την αλία και από τον τουρισμό που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να διατηρήσουμε το ζαχαροκάλαμο, τη ζάχαρη, την μπανάνα ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά. Έχουμε κάποια προβλήματα για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, γιατί ξέρετε ότι εμείς σε αυτά τα νησιά των υπερπόντιων περιοχών έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν έχουμε εκμεταλλεύσεις ε, ε μεγεθών σαν αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη. Ε, τι μπορούμε να έχουμε λοιπόν για να υπάρχει κάτι λοιπόν χρειάζεται απλοποίηση για τους μικρούς αυτούς γεωργού ε, απλοποίηση για το άρθρο 349 για τις ε, ενισχύσεις ε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι γεωργοί δεν μπορούν ε, να ε, έχουν αυτή την απλοποίηση, να υπάρχει αυτή η τεχνολογία επίσης. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Θα ήθελα να ξέρω τι μας προτείνετε για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι γεωργοί που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σήμερα θα μπορέσουν να επιβιάσουν. Τι μπορείτε να μας προτείνετε σήμερα κύριε Χόγκαν. Η κυρία Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις, τίποτα περισσότερο. Όταν αναφέρεστε ε, στο ένα δις, θα ήθελα να ξέρω Ποιες απαιτήσει θα πρέπει να πληρούν οι γεωργοί για να λάβουν τμήμα αυτών των χρημάτων. Και δεύτερη ερώτηση. Εάν ε, η Επιτροπή μας θα θεωρείς τους περιοχής ε, και το ρύζι και τα εσπεριδοειδή της Μεσογείου. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το, την ζάχαρη, τα, δημητριακά, τα σιτηρά και ε, το βόλιο κρέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ ενώπιον μας για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, η οποία κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική για να ξεκινήσουμε καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ των οίκων μας και να ε, ε, συμφωνήσουμε και ποιες προτεραιότητες έχουμε. Ξέρετε ότι σήμερα σας ζητούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες για την ΚΑΠ ε, και τη μεταρρύθμισή της. Ε, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί βεβαίως, αλλά πρέπει ε, να αναλάβουμε και τη δύσκολη πρόκληση να ανταποκριθούμε σε πολλά αιτήματα των πολιτών και των καταναλωτών και να υπάρχει σωστή φροντίδα για όσους ασκούν γεωργικά επαγγέλματα στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση την οποία θα ήθελα να ελπίζω ότι θα διαβάσετε εκεί που πρέπει. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ζητάμε από του γεωργού να κάνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντο, περισσότερα για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, περισσότερα για τον ε, διεθνή ανταγωνισμό και από την άλλη να κάνουμε περικοπέ στι ενισχύσει τη ΚΑΠ. Πιστεύω αντιθέτω ότι αν θέλουμε να προσφέρουμε μέσα αντίστοιχα των φιλοδοξιών μας θα πρέπει να δώσουμε νόημα σε αυτόν τον προπολογισμό για τη γεωργία και να στοχεύσουμε σε αυτούς που πραγματικά χρειάζονται χρήματα και να τους δώσουμε όχι μόνο γεωργική φιλοδοξία αλλά και διατροφική και περιβαλλοντική φιλοδοξία. Ο κύριο Αντέμουφ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τον σταθερό διάλογο που είχαμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής Γεωργίας. Εγώ εκπροσωπώ τη Βουλγαρία και είμαι μέλος του ΕΛΚΣ αυτήν την Επιτροπή. Και δεν, πρέπει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε ισότιμη με μεταχείριση των Ευρωπαίων Γεωργών και γι' αυτό υπάρχει μια σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων. Για αυτή, τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Επίσης, ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη και τι συνδεδεμένε ενισχύσει. Αυτές οι συνδεδεμένε ενισχύσει προασπίζουν συγκεκριμένα είδη παραδοσιακή παραγωγή και βοηθά τι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σκόπιμο λοιπόν να κρατήσουμε το ισχύον ε, επίπεδο συνδεδεμένων ενισχύσεων και ενδεχομένως να διαβρύνουμε και το πεδίο εφαρμογή τους. Δεύτερη ερώτηση για του μικροκαλλιεργητέ και τι μικρέ αγροτικέ εκμεταλλεύσει. Το απλοποιημένο καθεστώ για του μικροκαλλιεργητέ είναι ένα σωστό βήμα προ μια καλή κατεύθυνση. Τι άλλο όμω θα πρέπει να κάνουμε για να διευκολύνουμε του μικρού ευέλεια, μικρού κλίμακα να εφαρμόσουν και του ε, νέου περιβαλλοντικού στόχου τη ΚΑΠ. Επίσης, να αποκλείσουμε κάποιους μικρούς καλλιεργητές από την αιρεσιμότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τολγέ. Συγγνώμη, δεν έχω μάθει ακόμη όλα τα ονόματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την παρουσία σας και για την ομιλία σας. Ε, είπατε και τα θετικά και τα αρνητικά. Είμαι νέα Ευρωβουλευτής. Μία ερώτηση για τη διαφάνεια για τη διαδικασία, για τη σύναψη τη συμφωνία Μερκοσούρ. Έχουμε μελέτη αντικτύπου. Προβλέπετε να κάνετε τέτοια μελέτη. Και πότε θα μα τη στείλετε, εάν πρόκειται να την κάνετε. Γιατί αναφέρεστε σε αυτό το δι, ένα δι. Πώ θα μπορέσουμε να το διοχετεύσουμε στου γεωργού που θα το χρειαστούν. Πώ λοιπόν προβλέπετε να καθορίσετε τι διαδικασίε, Ποιοι θα έχουν ε, δικαίωμα σε αυτή τη χρηματοδότηση και από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά. Άλλο επίκαιρο θέμα. Ο Μπόρι Τζόνσον θα γίνει πρωθυπουργό. Θέλει να αποχωρήσει στι 31 Οκτωβρίου. Ακόμη και χωρί συμφωνία. Τι προβλέπετε για τον προβλησμό του 2020 για την κοινή γεωργική πολιτική σε περίπτωση αποχώρηση χωρί συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει Ο κύριο Ρίτσι. Η κυρία Ρίτσι. Κυρία Ρίτσι. Κυρία Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσία σας και για το ότι ήρθατε να μας μιλήσετε αλλά και να μας ακούσετε. Είμαι νέα τώρα, δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέροσταν, αναφέρεσταν ε, για στην, ε, στην ε, διαμάχη που είχατε με τον κύριο Φλάνναγκαν. Αλλά ελπίζω να πάτε καλύτερα, όπως θα πει και η χώρα σας αθλητικά. Αλλά με απογοήτευσε το ότι δεν είπατε τίποτα για την ανάπτυξη της Υπέθρου. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι η Επιτροπή μας εστιάζει κυρίως στη γεωργία. Αλλά εγώ είμαι εδώ γιατί ενδιαφέρομαι για την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη της Υπέθρου. Και κανεί εδώ μέσα μέχρι στιγμής, εκτός από την συνάλφο Μούλε, δεν αναφέρθηκε στο θέμα. Υπάρχουν πολλές εντάσεις ε, διαφορετικής φύσης. Για παράδειγμα, απερίμωση και ε, μόνο οι ηλικιωμένοι μένουν σε ορισμένε περιοχέ. Και αυτά πρέπει να τα κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σμιθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, χαιρόμαστε που σα ξαναβλέπουμε. Και χαίρομαι και, που, και εγώ που είμαι πάλι μέλος τη γιατί δεν ήμουν προηγουμένω. Θυμάμαι την ε, ακρόασή σα για την επιβεβαίωση, όπου συζητήσαμε αν, είναι σκοτσέζικα, αν τα σκοτσέζικα ή τα ιρλανδικά ουίσκι τα καλύτερα. Δεν νομίζω ότι καταλήξαμε, αλλά καλό που συνεχίζουμε το διάλογο. Και μετά από αυτά που είπε η κυρία Τολοέ για την αποχώρηση στις 31 Οκτωβρίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως είπα, θα δούμε. On verra. Τρεις ημερομηνίες του Brexit ε, ήδη ε, δεν υλοποίησαν τον Brexit. Γιατί καταφέραμε να τι αποτρέψουμε. Και εγώ, ω Σκοτσέζο Ευρωβουλευτή, η δουλειά μου είναι ε, να σταματήσουμε τον Brexit. Θεωρώ ότι η διατήρηση τη ενότητα και τη ακαιρεότητα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και λυπάμαι αν ορισμένοι στενοχωριούνται. Πολύ συγκεκριμένη ε, πρόταση που θα κάνω τώρα. Τα πήγατε πολύ καλά στη συζήτηση για τον Brexit και πρέπει να σα συγχαρώ. Χρειαζόμαστε μια υπηρεσία που να ε, ε, πολύ γρήγορα να μπορεί να διαψεύδει τα διάφορα ψεύδη που λέγονται για την γεωργική πολιτική. Ανοησίε λέει ο, ο Βρετανός Πρωθυπουργό για διάφορα υγειονομικά μέτρα και πρέπει αυτό να σας βοηθάει να ε, αντιμετωπίζετε την ε, παραπληροφόρηση για συμφωνίε ελευθερών εμπορίου όπως το Μερκοσούρ αλλά και άλλες. Αυτό θα σα βοηθούσε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ούπε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πριν από μία πενταετία, όταν ήσταν ακόμη υποψήφιος επίτροπος, σας ρώτησα στην ακρόαση που είχαμε οργανώσει τη γνώμη σας για τις άμεσες ενισχύσεις. Και είπα, είχατε υποσχεθεί ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να λύσετε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει καθόλου το ζήτημα των άμεσων ενισχύσεων και σε μερικές χώρες ε, οι γεωργοί λαμβάνουν το 65% των ενισχύσεων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα λοιπόν στις άμεσες ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν λύσουν αυτό το πρόβλημα θα εξακολουθεί να είναι διχασμένη η Ευρώπη σε Ευρώπη παλιών και νέων χωρομελών, σε γεωργούς πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο δυνατόν να επιληθεί το ζήτημα της άνησης ε, κατανομής των άμεσων ενισχύσεων. Επίσης, πολλές φορές μιλάμε για, για τα θέματα των τιμών, της τιμής αγοράς ή της προστασίας των γεωργών που προσφέρουν ε, πρώτες ύλες. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη για το Μερκοσούρ. Τι θα γίνει με τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Είπατε ότι θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικό και με τι αγωγέ και για τι αγωγέ να τηρούνται και θα ελέγξετε. Ε, κοιτάξτε. Δυσκολεύω να το πιστέψω. Πώς θα το ελέγξετε. Διότι θα πρέπει να δεχθούν οι χώρες Μερκοσούρ τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ξέρετε ότι είμαι ενθουσιοδός υπέρ της ε, μεταβατικής περίοδου. Λέτε ότι προβλέπετε μια τέτοια μεταβατική περίοδο. Ε, πρόκειται για τον πρώτο πυλώνα που θέλει ενίσχυση για να υπάρξει ασφάλεια για τις ε, εργασίες αυτές. Πείτε μας ακριβώς το κάνετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω. Με προβληματίζει όμως το μέλλον της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόβλημα δεν έχουν μόνο οι γεωργοί. Και σε άλλους τομείς αλλάζουν οι πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνται προβλήματα. Πώς μπορούμε όμως να πετούμε όλο και περισσότερα από τους Ευρωπαίους γεωργούς δίνοντάς τους λιγότερα κονδύλια χαμηλότερα κονδύλια. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ενισχύσεων μεταξύ ανατολικών και δυτικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην πραγματικότητα δεν αμείβουμε επαρκώς τους Γιώργους για το έργο που επιτελούν. Περνάω τώρα στο Μερκοσούρ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς θεωρείτε θετική τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ. Εδώ όμως έχω τη γνώμη των ε, άμεσα ενδιαφερομένων που προβληματίζονται για την ε, εισρωή εισαγόμενων προϊόντων που δεν θα τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ο κύριος Τσερουσό, καλημέρα. Τζαρούσο. Κύριε Επιτροπέ, οι χώρες της Μερκοσούρ δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τα εργασιακά, περιβαλλοντικά και λοιπά πρότυπα για την προστασία των ζώων. Πώς θα παρακολουθήσουμε όμως αυτή την πρόοδο, διότι το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης προβλέπει αναστολή της συμφωνίας εάν δεν αυξηθούν αυτά τα πρότυπα. Ε, διαπιστώνω με ανησυχία ότι ο κύριος Μπολσονάρο αποφάσισε να εγκρίνει 150 φυτοφάρμακα στην εθνική του νομοθεσία. Πώς θα διαχειριστούμε λοιπόν ε, την ε, ε, εισαγωγή από χώρες που χρησιμοποιούν τέτοια φυτοφάρμακα και τι γίνεται με την αρχή της προφύλαξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, επειδή έχουμε προβλέψει ένα δις ευρώ για μέτρα προστασίας των γεωργών, θα θέλαμε να ξέρουμε με ποιο τρόπο σκοπεύετε να διοχετεύσετε τα, τα χρήματα και πώς θα κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ακούω τον Επίτροπο να αναφέρει θέματα τόσο σημαντικά όσο η γεωργία, ε, είμαι ανάμεσα στην ανησυχία και το δέος σε τι χρησιμεύει η γεωργία. Χρησιμεύει για να τρέφουμε τους πολίτες μας και ε, είναι πολύ σημαντικά τόσα γίνονται από αυτού και επομένω πρέπει να γίνει η συζήτηση της βιοργίας σε πραγματική συζήτηση για την κοινωνία. Για παράδειγμα, τα φυτοφάρμακα. Η σχέση μεταξύ υγείας και φυτοφαρμάκων είναι πολύ σημαντική και πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς να μεταβούν σε μια γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα. Όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, ο, ο ρόλος της γεωργίας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ε, σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση και με τα φυτοφάρμακα, Επομένω, θα πρέπει να βοηθήσουμε τη γεωργία να προστατεύσει τη βιοπικιλότητα που είναι προ όφελο τη γεωργία και τη γεωργική παραγωγή. Για το κλίμα, σχεδόν το έχετε υποβεβαιώσει στι μεταφορέ ε, των ζώων. Ε, ο Γεωργός έχει μεγάλη σχέση με την κλιματική αλλαγή γιατί εκπέμπει ε, άρια του φαινομένου της θερμοκηπίας, πλήττεται και από την ξηρασία, αλλά η λύση για την κλιματική αλλαγή είναι να υπάρχει καινοτομία όπω είναι η αγροοικολογία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πραγματική συζήτηση για την κοινωνία, θα πρέπει να υπάρχουν θέσει εργασία για τη γεωργία, να εγγυηθούμε το εισόδημα των γεωργών και να ε, λάβουμε υπόψη του γεωργούς και του καταναλωτές και τότε θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε και επιπλέον προπολογισμού για να υποστηρίξουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η γεωργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να μην ε, υπερβαίνει το χρόνο σας. Η κυρία Βίλαν. Χαίρετε και εγώ με νέο μέλος και ήρθα σε αυτή την Επιτροπή λόγω των ε, υπαρξιακών απειλών που υφίσταται το πλανήτη μας. Είμαι γεωργός και είμαι πολύ απογοητευμένη. Συζητάμε για μικροπράγματα και διακοσμητικές αλλαγές. Δεν ασχολούμεθα με τα βασικά θέματα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ε, ε, μία αγορά κρέατος που να είναι διαφανής και οικολογικά ε, συμβατεί με τη λειτουργία της. Ρωτάω λοιπόν, τι θα γίνει τώρα λοιπόν που έχουμε επανεθνικοποίηση. Πώς ακριβώς θα ελέγξετε λοιπόν τα εθνικά σχέδια αν δεν έχουμε ε, αντικειμενικούς δείκτες. Για παράδειγμα, στον πρώτο πυλώνα της κοινή γεωρικής πολιτικής θεωρούνται μέτρα που βοηθούν το περιβάλλον, να βελτιώνουμε, μάλλον καλύτερα, να κάνουμε πιο εντατική γεωργία μέσω εισαγωγής φίλτρων που μειώνουν τις εκπομπές ε, κακών αερίων. Μα αυτό δεν είναι προστασία του κλίματος. Στην ουσία είναι μασκάρεμα. Πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτή τη θητεία, διότι αλλιώς δεν θα υπάρξουμε ούτε εμείς, ούτε οι επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γούσεν. Ευχαριστώ. Όχι μόνο κάνει ζέστη, αλλά υπάρχει και μεγάλη ξηρασία, ιδιαίτερα στην Ολλανδία. Αναλάβατε κάποιες δράσεις για να ε, αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και θα χρειαστεί και φέτος κάτι παρόμοιο τι θα κάνετε, θα υπάρξουν κάποιοι κανόνες ε, κατάλληλοι. Δεύτερον, το μποϊκό των ρωσικών προϊόντων. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο συζήτησα με διάφορους ε, παραγωγούς που θίγονται ιδιαίτερα από αυτό το μποϊκότ. Οπότε, τι μέτρα θα λάβετε ούτω ώστε ο τομέα των ε, φρούτων και λαχανικών να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά το Mercosur, Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Πολύ καλά να κάνουμε εμπορικές συμφωνίες, αλλά θα πρέπει τα προϊόντα που εισάγουμε να συμμορφούνται με κανόνες και για την ε, φυτογεωνομική κατάστασή τους και για την ευημερία των ζώων. Θέλουμε περισσότερες εξηγήσεις για αυτά τα θέματα. κυρία Σμιτ Μπάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι νέα βουλευτής από την Αυστρία. Οι γεωργοί μας έχουν ανησυχίες. Και ανησυχούν ιδιαίτερα λοιπόν όπως σας είπα γιατί έχουν θυγεί. Γιατί και εγώ είμαι γεωργός και ξέρω τις ε, προκλήσεις και τις απαιτήσει που μας επιβάλλουν οι ίδιοι καταναλωτές. Το άνοιγμα των αγορών με προϊόντα πολύ χαμηλότερων προδιαγραφών από αυτά στα οποία είμαστε συνηθισμένη, και οι περικοπέ τη κοινή γεωργική πολιτική είναι ακατανόητο όλα αυτά. Γι' αυτό, ερώτηση, προτίθεται η Κομισιόν να κάνει μια μελέτη για τι συγκεκριμένε επιπτώσει αναχώρα και αναευαίσθητο γεωργικό τομέα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη πιο υπεύθυνα. Και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικέ ειδικέ ανταγωνισμού. Αναφέρθηκαν ορισμένα τέτοια θέματα. Κόστο παραγωγή, προδιαγραφέ, βιώσιμη τρόπη παραγωγή και φυσικά και η ευημερία των ζώων. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τη γεωργία αλλά και για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπούσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από ό,τι λένε οι ερευνητέ, μας μένουν 11 χρόνια αν είναι να αποτρέψουμε την ε, κατάρρευση του κλίματος. Οι νέοι ανακατομμύρια διαδηλώνουν. Αλλά ο, ο κύριος Μπολσονάρο δεν ενδιαφέρεται. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, καταστρέφονται τα μεγαλύτερα τροπικά βροχοδάση. Τον περασμένο Ιούνιο καταστράφησαν 750 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι περίπου η διαστάση του Αμβούργου και ε, αναχρόνω θα καταστρέφονται 60% παραπάνω εκτάσεις ε, τρόπο δάσους. Για να φτιάξουν καλλιεργήσιμες ε, εκτάσεις, για να παράγουν ζωοτροφές με τις οποίες θα εξάγουν σε τιμές dumping κυρίως προς τις Ηνωμένε Πολιτείε και στην ε, Ευρώπη. Και η κτηνοτροφία σημαίνει τεράστια παραγωγή μεθανίου που είναι πολύ βλαβερότερο από το δεξίδιο του άνθρακος. Πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις λένε να παγώσει αυτή η συμφωνία. Αλλά ο ακροδεξιός Μπολσονάρο θέλει να συνεχίσει την ε, ακραία πολιτική του. Και αυτά, όπω ξέρετε, είναι και κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των περιβαλλοντικών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόγκ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του. Θα ήθελα και εγώ ως νέα να συμφωνήσω με τον Άλ Σμιτ Μακάρι να μην είμαστε μόνο νέα μέλη, αλλά και μακρόβια μέλη αυτής της Επιτροπής και να μην υλοποιηθεί το Brexit στις 31 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τον ιδιαίτερα ολοκληρωμένο χαρακτήρα που έχει η Γεωργία και η παραγωγή τροφίμων στην Ιρλανδία, <clears throat> τι μέτρα θα λάβετε ώστε σε περίπτωση Brexit να Συνεχιστεί πρόσβαση και μετά το Brexit ε, σε κατάλληλη συσκευασία μεταποίηση των προϊόντων ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε σπάνι τροφίμων στην δύσκολη μεταβατική περίοδο. Και σε ό,τι αφορά το Mercosur και άλλοι αναφέρθηκαν ε, στις περιβαλλοντικές ανησυχίες που εγείρει. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στη Βόρεια Βερλανδία ένα ε, κιλό βοήου παράγει 60 κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Ενώ στις, ε, στο, στην Νότια Αφρική έχουμε πολύ μεγαλύτερη ε, έκρηση τέτοιων αέριων, αέριων του θερμοκηπίου. Θα είναι τεράστιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα δηλαδή με τέτοιε παραγωγή και με ολέθριε συνέπειε για τι κλιματικέ αλλαγέ και την υπερθέρμανση του πλανήτη, αν δεν δούμε τι συμφωνίε αυτέ με το πραγματικό του πρόσωπο. Ωραία. Μίλησαν όλοι. Όσοι ήταν στο κατάλογο 33 συγκεκριμένα. Ο Επίτροπος έγραφε μανιωδό. Αλλά θα είναι δύσκολο να απαντήσει αναλυτικά σε όλε τις ερωτήσεις. Θα ήταν δυνατόν σε 10 λεπτά, κύριε Επίτροπε, να έχουμε κλείσει τη συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα βάλω τα δυνατά μου. Καταρχήν, συμφωνία με τη... τις χώρες Μερκοσούρ. Μερικοί κατάγεστε από χώρες που ε, είστε υπέρμαχοι του Μερκοσούρ γιατί βγήκατε κερδισμένοι από τα θέματα τα βιομηχανικά των δημόσιων ε, συμβάσεων και άλλοι όπως η Γερμανία και η Γαλλία είστε κατά λόγω της γεωργίας. Αλλά και άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία τάχθηκαν υπέρ κάποιων τυχών του Μερκοσούρ και ε, υπέρ της συμφωνίας ανάλογα με τον τομέα που ευνοείται. Ε, άλλοι τομεί βρέθηκαν πολύ πιο ευνοημένοι, η γεωργία ίσως λιγότερο. Εμείς προσπαθήσαμε να μετριάσουμε τις παραχωρήσεις που χρειάστηκε να κάνουμε στη γεωργία. Και αν έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ παραχωρήσεων που κάναμε στους μη γεωργικούς τομείς, που επιτύχαμε συγγνώμη στους μη γεωργικούς τομείς, θα πρέπει κάποιες υποχωρήσεις να γίνουν στο γεωργικό κλάδο. Πάντως πρόκειται για μια συμφωνία 88 δισεκατομμύριων ευρώ. 760 εκατομμύρια άνθρωποι εμπλέκονται. Και θα πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα του συνόλου των κλάδων. Συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει μελέτη αντικτύπου για κάθε τομέα ξεχωριστά για να δει πώ η συμφωνία θα επηρεάσει τον κάθε τομέα. Αυτό γίνεται συνήθω ε, και για όλε τι συμφωνίε. Εδώ έχουμε όμω, αν δούμε τις δασμολογικές, ε, τους δασμούς που καταργήθηκαν και αν το δούμε διακλαδικά αυτό, βλέπουμε ότι έχουμε καθαρά 4,5 δισεκατομμύρια δασμούς που καταργήθηκαν αυτό δεν έχει στόχο να υποτιμήσει τις υποχωρήσεις που κάναμε στη Γεωργία. Σίγουρα χρειάστηκε να γίνουν 45 δισεκατομμύρια στα αγαθά, 23 ε, δισεκατομμύρια στις, ε, στις υπηρεσίες. Είναι τίμα της συμφωνίας. Και οι πρωθυπουργοί στο χωρό, το χωρό σας, οι πρωθυπουργοί, οι πράσινοι θα είναι ε, κυβέρνηση σύντομα και είχατε, ε, ε, μπορεί να είναι σύντομα στο σχηματισμό της κυβέρνησης, αλλά κάνατε πολλές υποσχέσεις. Σκεφτείτε όμως τι θα γίνει αν βγείτε τελικά. Θα πρέπει να προσέξετε τι επιθυμείτε και τι εύχεστε. Εσείς είστε στη, στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Μακάρι να ήσασταν. Καλύτερα να επικεντρωθείτε στο Brexit, κύριε Κάρθη, γιατί είστε 7 μέλη Το έχω πει πολλές φορές, ε, επανειλημμένως. Είστε 7 Ευρωβουλ... Ε, είστε 7 ε, από τη Βουλή των Κοινοτήτων και θα μπορούσατε να κάνετε πραγματικά τη, διαφορά, να φροντίσετε να αποτραπεί το Brexit. Και φαντάζομαι όσοι αναφέρθηκα στο Brexit και τη Γεωργία να γνωρίζουν τις δυσκολίες που γίνεται. So Δυστυχώς μιλούν ταυτόχρονα και οι δύο μιλητές. Μακάρι να πείσετε τους συναδέλφους σας και να κατεβείτε από τα ύψη στα οποία στέκεστε και να δώσετε μάχη ώστε να παραμείνει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ο μόνος τομέας άλλωστε που έχουμε προβλήματα. Κύριε Κάρθη, το 2004, λίγο πριν ίσως <laughs> από εσάς, 170.000 τόνοι βόλιο ήταν επιτάπητος, απορρίφθηκαν από τη Βραζιλία και το μειώσαμε αισθητά αυτό το ποσό. Η κυρία Μαγκίνε έκανε πιο σε ερωτήσει. Τι θα γίνει σήμερα με την κρίση του βοηού κρέατος. Εσείς για πέντε χρόνια μιλούσατε για τις, για τις ψήφους και είπατε ότι έχετε περισσότερες. Κι όμως ε, η, η δική της ε, ιδιότητα και το δικό της αξίωμα είναι υψηλότερο από το δικό σας. Και ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να θέσουμε το Brexit στο πλαίσιο, σε ευρύτερο πλαίσιο και υπό το πρίσμα του Μερκοσούρ. Και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να δρούμε όπως δρούμε, γιατί με ρωτήσατε για τα περιβαλλοντικά θέματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, αν εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προσπαθήσει να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες του κόσμου. για ανεξάρτητες ε, συμφωνίες. Και αν συνάψει συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ, τι προδιαγραφές και πρότυπα θα έχουν ε, τα εισαγόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο προϊόντα από το Μερκοσούρ μετά το Brexit. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό για πολλούς και ευαίσθητους κλάδους, Γεωργία και άλλους. Και με μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που θα συνάψουμε το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση Brexit, σε περίπτωση αποχώρηση. τα βρετανικά προϊόντα θα πρέπει να τηρούν τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που διαπραγματευθήκαμε με το Μερκοσούρ, σε περίπτωση που ε, συμφωνήσει ξεχωριστά με το Μερκοσούρ. Και πολύ φαίνεται ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι η πατρίδα σας ε, είναι ε, αρμόδια για την διενέργεια των ελέγχων και την τήρηση των προδιαγραφών και των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα γίνει αστυνόμευση, εθνικό επίπεδο ε, για την τήρηση των προδιαγραφών. Και αν δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι σε κάθε χώρα, θα πρέπει αυτό να το δει το κάθε κράτο χωριστά. Και έγιναν όντω, κύριε Αντρία, κάποια σκάνδαλα στο παρελθόν με τα πουλερικά και τα πουλερικά που εισάγονται στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 100.000 ε, τόνους γιατί έχουν βελτιωθεί οι έλεγχοι και μάλιστα συνεργαζόμαστε με τη Γαλλία να το, να το επιτύχουμε. Το 2017 είχαμε 100.000 τόνους λιγότερους και το 2018 μάλλον σε σχέση με την κρίση που είχαμε το 2017 για τα πουλερικά. Χρειάζονται λοιπόν αυστηρή έλεγχη αλλά κανένα προϊόν δεν θα ε, δεν θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μερκοσούρ με 100% έλεγχους. Και μάλιστα είχαμε πριν από 2-3 χρόνια ένα σκάνδαλο πάλι με κρέας. Σίγουρα ε, το ζήτημα της τιμής του βοηού κρέατος είναι σημαντικό για τους κτηνοτρόφους. Και εμείς συμφωνήσαμε 100 ε, εκατομμύρια ευρώ να δοθούν σε ένα μόνο κράτος και μάλιστα οι υπόλοιπες χώρες συμφώνησαν με αυτό. Και σίγουρα ε, θα πρέπει να ε, δείξει ευγνωμοσύνη η Γεωργία και να ευχαριστήσει. Εγώ το, το διαπίστωσα γιατί κανένας, κανένας άλλος Ευρωπαίος δεν καταψήφισε αυτή την πρόταση για να δοθούν αυτές οι ενισχύσεις στους Ιρλανδούς κτηνοτρόφους. Ήταν ομόφωνη η απόφαση και θα πρέπει να δείξουμε την αναγνώρισή μας και την εκτίμησή μας γι' αυτό και την αλληλεγγύη που έδωσαν οι υπόλοιποι. Τώρα, θα πρέπει να δούμε πώς γίνονται οι δουλειές και οι η έλεγχη στα κράτη-μέλη και δεν ξέρω και τη δική μου. Και να το δούμε για τα ευαίσθητα προϊόντα. Αυτό το κάνουμε στην Ισπανία. Υπήρχαν προβλήματα με τα σπεριδοειδή, με τι επιτραπέζιε ελιέ. Και στην Πολωνία έχουμε πρόβλημα ξηρασία. Και 7 χώρε και η Γαλλία μεταξύ του ζήτησαν προκαταβολέ 70% ε, ε, σε σχέση με το 50% που είχαμε μέχρι στιγμής. Και Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την ανάγκη ρευστών που έχουν οι γεωργοί, θα εξετάσουμε θετικά αυτά τα αιτήματα. Και θα ήθελα να πω στην Γαλλίδα Ευρωβουλευτή, όντως εξετάζουμε πολύ θετικά το αίτημα της Γαλλίας για την αύξηση του ποσοστού προκαταβολής και μάλιστα και άλλες έξι χώρες, η Πολωνία μεταξύ άλλων που ζήτησαν ε, τέτοιες προκαταβολές, μάλλον θα τις λάβουν κυρία Χάζεκαπ έθεσε κάτι για τη Ρουμανία. Δεν το γνωρίζω. Ε, όντως το θίξατε και στον κύριο Αντρουκάητης. Δεν γνωρίζω ε, το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί εκφεύγει των δικών μου αρμοδιοτήτων. Πάντως θα το θέσω και στο συνάδελφο Αντρουκάητης και θα λάβετε διεξοδικές εξηγήσεις. Συμφωνώ με όσου θέλουν πλήρη χρηματοδότηση τη ΚΑΠ και θα συνεργαστούμε με εσά και τα κράτη-μέλη για να το πετύχουμε. Αλλά τέσσερι χώρε δεν θέλουν να αυξηθεί ο γεωρικό προπολογισμό ε, ή ο κοινοτικό προπολογισμό λόγω Brexit που δημιουργεί ένα χρηματοδοτικό κενό 12 δισεκατομμυρίων. Οπότε, χωρί χρήματα δεν μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση και να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων. Κάποιοι πρωθυπουργοί είπαν ότι θέλουν περισσότερα κονδύλια για τη μετανάστευση, ε, την άμυνα, την ασφάλεια, άλλοι για την τεχνολογία και την έρευνα. Ωραία όλα αυτά και ε, σωστή στόχη, αλλά θέλουμε και κονδύλια για να υλοποιηθούν οι πολιτικέ. Πάντω, συνεργαζόμαστε με όλε τι κυβερνήσει για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κυρία Νόιχλ, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο για το τι είπε στην ομιλία τη η κυρία Φοντερ Λάιεν. Δεν είναι η την πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσιώπησε το θέμα της Γεωργίας και το γνωρίζω αυτό εκ των έσω. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, των άμεσων ενισχύσεων, μείζον ζήτημα για χώρες Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως για τις Βαλτικές χώρες, αυτό όντως ήταν ε, ζήτημα της μεταρρύθμισης του 2013 και του προϋπολογισμού του 2013. Εμείς είπαμε να πάμε στο μισό της πρότασης. Όχι στο 100% σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων, αλλά τουλάχιστον να βρεθούμε κάπου στη μέση, στο 50%. Και αν υπάρξουν επαρκή κονδύλια και αποφασίσουν οι Πρωθυπουργοί να εξασφαλιστεί η ισότητα των άμεσων ενισχύσεων, φυσικά συμφωνώ. Είμαι υπέρ της πλήρους σύγκλησης των γεωργικών ενισχύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μερικές χώρες επικεντρώνονται στα κριτήρια για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων. Στις γεωπονικές συνθήκες, ε, το, την τιμή της ε, γης, των αγροτεμαχίων. Πάντως εγώ είμαι υπέρ ε, της ισότητας των άμεσων ενισχύσεων, αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος, μόνο μία φωνή. Αυτό θα το αποφασίσουν οι χώρες και στα πλαίσια του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Πολλοί αναφερθήκατε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρώτη φορά έχουμε... Ε, προκαθορίσει τέτοιο αποθεματικό για ένα τομέα σε περίπτωση διαταραχής αγοράς. Και είχαμε και από το ρωσικό εμπάρκο τέτοια εμπειρία διαταραχής αγοράς. Εκεί αφιερώσαμε 1,7 δις επιπλέον του γεωργικού προϋπολογισμού που είχε αποφασιστεί το 2013-2014. Οπότε τα χρήματα αυτά α, αναγγέλθηκαν σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καθησυχαστεί η γεωργική κοινότητα γιατί υπάρχουν πολλές ανησυχίες στους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Θελήσαμε να τους καθησυχάσουμε ότι αν πραγματοποιηθεί το απευταίο θα υπάρχουν μηχανισμοί σε περίπτωση διαταραχής με τις 99.000 τόνους βοήου που θα εισέλθουν στην αγορά. Και επιπλέον θα λάβουμε υπόψη και το θέμα των πουλερικών. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους γεωργούς μας όπως μπορούμε. Και το 1 δισεκατομμύριο είναι ένα μήνυμα προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν λάβει χώρα διαταραχή ή στρέβλωση αγορά, θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια. Σε περίπτωση μόνο όμω που υπάρχει τέτοια διαταραχή. Και στο παρελθόν είχαμε κριτήρια για να το λάβουμε υπόψη. Η κυρία Πύρικ μίλησε για το μοσχαρίσιο κρέα και αν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία ή γίνεται διάκριση μεταξύ βόηου κρέατο και μοσχαρίσιου ή άλλων προϊόντων. Όχι. Ε, για τα πουλερικά είχαμε 80.000 τόνους και αυτό είναι ένα μικρό των 14 εκατομμυρίων εσωτερικής κατανάλωσης και θα μπορούσαμε η αγορά να φτάσει ε, στους 223.000 τόνους το χρόνο. Ήταν μία υποχώρηση, δεν μας αρέσει να κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά λάβαμε υπόψη την κατανάλωση στο βόλιο που μειώνεται, ενώ υπάρχει μια αύξηση στην κατανάλωση πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταβατικός κανονισμός, το έχω αναφέρει ήδη και πολύ το επαναλάβατε. αν συνεργαστούμε και καταλήξουμε σε αποτέλεσμα, θα τα καταφέρουμε. Πάντως είμαστε έτοιμοι. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουμε το ρυθμό που θα θέλαμε, θα φροντίσουμε να προασπίσουμε παρόλα αυτά στη μεταβατική περίοδο το γεωργικό εισόδημα. Και στην πρόταση της ΚΑΠ υπάρχει μια αλλαγή στους τομεακές ενισχύσεις στα πλαίσια του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς και για πρώτη φορά έχουμε κλαδική υποστήριξη, τομεακή υποστήριξη σε όλου του και όχι μόνο στα προκυπευτικά. Κάποιο από τη Βουλγαρία και άλλοι αναφέρθηκαν στου μικροκαλλιεργητέ. Εμεί προτείναμε ανώτατα όρια για να απελευθερωθούν ε, τα κονδύλια και για του μικροκαλλιεργητέ. Αλλά η Βουλγαρία ήταν κατά. Δεν θέλετε να φέρουμε από του μεγαλοκαλλιεργητέ για να δίνουμε στους μικρού. Οπότε από κάπου θα πρέπει να βρούμε τα κονδύλια. Αν εξοικονομήσουμε λοιπόν κάποια χρήματα από τα ανώτατα όρια, μπορούμε να ε, χρηματοδοτήσουμε τους μικροκαλλιεργητές. Ε, ίσως οι μεγάλοι γεωργοί να δυσαρεστηθούν, αλλά στην Βουλγαρία είναι περισσότεροι μικροκαλλιεργητές, όπως και στη Ρουμανία. Χρειάζεται πάντως πολιτική βούληση για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Τώρα, για το θέμα των προδιαγραφών και των Μερκοσούρ. Θέλω να το επαναλάβω και πάλι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και μεγάλη εξασφάλιση προς τους γιοργούς. Όλοι οι πόροι που είναι διαθέσιμοι με τη βοήθεια των κρατών μελών ώστε να έχουμε 100% ελέγχου ε, και ε, παρακολούθηση θα εφαρμοστούν. Αν χρειάζεται οποιαδήποτε εξασφάλιση ε, είμαι στη διάθεσή σα. Τώρα, για τα προϊόντα και τα όσα είπε η φίλη μας από τη Γουαδελόπη και τη Μαρτινίκα ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό. Θα διατηρήσουμε το συγκεκριμένο καθεστώς για το ΠΟΣΕΙ και τις ενισχύσεις που έχουμε για αυτές τις νησιωτικές χώρες που εκπροσωπείται. Δεν θα αλλάξει ε, κάτι. Προστατεύσαμε τον προπολογισμό τους και προστατεύσαμε και τις ε, συνθήκες εμπορίου που, που ισχύουν σήμερα θα ισχύουν ακόμα για τις υπερπόντιες περιοχές και τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Κύριε Λεμπρετών, δεν είπα ότι θα αρχίσουμε ε, να θυσιάζουμε το βόλιο κρέας για τον ίνο. Ε, μπορείτε να στρεβλώνετε αυτά που λέω, αλλά θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν έγινε καμία θυσία σε γεωργικό προϊόν. Δεν σας άκουσα να αναφέρετε τον ίνο ή και τα άλλα προϊόντα, στα οποία λάβαμε πολύ μεγάλα ε, στοιχεία και επιτυχία και γεωγραφικές ενδείξεις για πολλά προϊόντα, πολύ πλούσια προϊόντα από τη Γαλλία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολα. Ε, η σαμπάνια, για παράδειγμα, πολύ δύσκολο ε, να καταφέρουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιτύχαμε. Δεν ε, θυσιάσαμε κανένα τομέα για άλλους τομείς. Ο βιομηχανικός τομέας όμως στη Γαλλία επωφελείται πολύ από αυτή τη ε, συμφωνία. Σίγουρα ο γεωργικός τομέας πιέστηκε, αλλά υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Ο μηχανισμός, ε, όπως ζήτησαν οι Γάλλοι ε, για δικλείδες ασφαλείας με δασμούς και ποσοστώσεις που χρησιμοποίησαμε και στο παρελθόν. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν τα είχαμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Το χρησιμοποίησαμε το μηχανισμό αυτό στην Ιταλία για εισαγωγές από την Καμπότζη. Επομένως, μην θεωρείτε είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει προ όφελο ε, των Ιταλών ε, οριζοπαραγωγών και θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον, ε, αν χρειαστεί. καταφέραμε να το έχουμε στη συμφωνία και το πετύχαμε στη συμφωνία για το Μερκοσούρ. Κυρία Τολερέ, είχαμε πολλά ε, πράγματα. Η κυρία Μάλστρομ έχει έρθει πολλέ φορέ στο Κοινοβούλιο για να συζητήσει την εμπορική πολιτική. Έχει συναντηθεί με όλου του ενδιαφερομένους για το τι θα πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι η πιο διαφανή συμφωνία που έχει γίνει με όλου του ενδιαφερομένου και του εκπροσώπου κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει και μια δήλωση από το 2016 που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πολλέ συμφωνίε που έγιναν για την ανάπτυξη τη υπαίθρου σε αυτή τη διάσκεψη περιλαμβάνονται στην πρόταση τη ΚΑΠ. Το γεγονό ότι δεν ανέφερα σήμερα την ανάπτυξη τη υπαίθρου δεν σημαίνει ότι δεν μα ενδιαφέρει το θέμα. Και όσον αφορά το Ιρλανδικό και το Σκοτσέζικο ουίσκι, μπορούμε να κάνουμε και δοκιμασία, μα θέλετε να δείτε, να ελέγχετε και το προϊόν. Εμείς όμως έχουμε μια Ιρλανδική γεωγραφική ένδειξη και όταν θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω και το Σκοτσέζικο ουίσκι να μπορεί να αναγνωρίζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αυτό θα είναι τεράστια πρόκληση για το Σκοτσέζικο ουίσκι και να δούμε πώς θα επιληθεί. Αν η Βρετανική κυβέρνηση δεν προστατεύσει, ε, όπως για παράδειγμα με τις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, τότε σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα ε, και εκεί θα έρθει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει αν χρειαστεί. Ε, κύριε Πρόεδρε, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχω απαντήσει σε όλα. Κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω αφορά την ΑΕΟ Μιλάν και να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το να μην υπάρξει συμφωνία και αποχώρηση είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε σε θέση φυσικά να συζητήσουμε τώρα, γιατί εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επί της βάσης ότι θα υπάρξει συμφωνία. Ε, και συζητούσαμε και πριν από τις 29 Μαρτίου και μετά ε, ε, υπάρχουν μέτρα από το Μάιο του 2019. Υπάρχει χρηματοοικονομική στήριξη, αν υπάρξει κράχ ε, ή υπά, δεν υπάρξει συμφωνία και αποχωρήσει έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει η δεν υπαρξει συμφωνια και αποχωρησει ετσι το ηνωμενο βασιλειο υπαρχει η δυνατοτητα ε, συζήτησης λύσης για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες ε, συμφωνίες. Πρέπει να εξετάσουμε και το χειρότερο ενδεχόμενο. Ελπίζουμε να μην συμβεί, αλλά υπάρχει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης και ε, σχέδιο αναδίπλωσης. Και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει και στα σκαριά 16 νομοθετήματα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τέλος, να πω στον κύριο Μπούντα ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα ε, τα οποία μπόρεσαν να λάβουν τα κράτη-μέλη στο παρελθόν. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, για τη διασυνοριακή βοήθεια. Αυτό είναι τμήμα των συζητήσεων για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό μπορεί να έρθει και με την ε, συνδεδεμένη στήριξη και να συζητηθούν αυτά για να προστατεύσουμε τους διαφόρους τομείς. Πέραν της ε, κλαδική στήριξη που προσφέρεται για όλου του τομεί που δεν είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί που μπορούμε να συζητήσουμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία και να καθησυχάσουμε του αγρότε κυρίω στη Ρουμανία. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, αλλά ο Επίτροπος ε, δεν απάντησε για το ελαιόλαδο και τις χαμηλές τιμές ε, που ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Δεν θα ήθελα να μην απαντήσετε. Η πρόταση που σας ναι, η Ισπανική κυβέρνηση και ο κλάδος θα γίνουν αποδεκτές. Και κύριος ήθελα να πολύ σύντομα παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ο διάλογος περαιτέρω. Ευχαριστώ. Μια παρατήρηση επί της ουσίας. Πολλά από τα ερωτήματά μας είπατε ότι τα προβλήματα οφείλονται στις αποφάσεις των κρατών μελών. Και επειδή θα σας βρούμε μερικές εβδομάδες ε, για τις ακροάσεις, από τη Λισαβόνα και μετά είμαστε στις νομοθέτες. Είμαστε σοβαροί εμπλεκόμενοι. Πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη. Και εμείς θα το λάβουμε υπόψη δεν υπάρχει μόνο το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και εμείς παίζουμε πλήρως το ρόλο μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα νομίζω ότι αναφέρθηκα τουλάχιστον 10 φορές στους συνομοθέτες. Με εκπλήσει που εξακολουθείτε να ανησυχείτε. Έχω την μέγιστη δυνατή, το μέγιστο δυνατό συμβασμό για το Κοινοβούλιο. Εγώ έρχομαι τακτικά εδώ, δεν χρειάζεται να με υπενθυμίσετε τη σημασία του Κοινοβουλίου πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιοι άλλοι στο παρελθόν. Συμμερίζομαι πλήρω. Αυτό που σα είπα είναι ότι εγώ προσπαθώ επικοδομητικά με την Επιτροπή σα να διασφαλίσω την πλήρη χρηματοδότηση τη κοινή γεωργική πολιτική. Είναι ο κοινό μα στόχο. Τώρα μην αρχίσουμε τώρα σημειολογικέ ε, συζητήσει για το θεσμικό θέμα. Τώρα για το ελαιόλαδο. Ο κύριο Πλάνα και η κυρία Αγγιλέρα ε, με πλησίασαν για το θέμα αυτό, το εξετάζουμε τώρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον τομέα του ελαιολάδου. Δεν έχω απάντηση σήμερα. Ε, αξιολογούμε την κατάσταση και ελπίζω να μπορέσω να σα απαντήσω μέσα στι επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ο κύριος Επίτροπος είπε ότι κάποιες ερωτήσεις ε, που δεν απαντήθηκαν θα απαντηθούν από τις υπηρεσίες του τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε, πολύ χρόνο, σήμερα το απόγευμα και φυσικά θα υλοποιήσουμε την προσφορά που μας κάνετε για περαιτέρω συνεργασία. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποχωρήσετε κύριε Επιτρόπη για σήμερα και μετά λοιπόν μια σύντομη διακοπή. Θα συνεχίσουμε με τα επόμενα θέματα της ημέρης διάταξης. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle, die jetzt anderes zu tun haben. Κοιτάξτε, αν έχετε άλλη δουλειά και δεν θέλετε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση για τον προπολογισμό, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Ich würde gerne in der Tagesordnung fortfahren. Λοιπόν, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην μέση διάταξη. Οπότε παρακαλώ, όσους ενδιαφέρονταν μόνο για τον Επίτροπο και όχι για τον προπολογισμό, τι σίγουρα ενδιαφέρουσε ε, κατηδίαν συζητήσεις, να τις εξαγάγουν εκτός εθούσης. Για να προχωρήσουμε. Έχουμε τώρα το σημείο 7. Γενικός προπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020. Λοιπόν, να σας τα διαβάσω αγγλικά έτσι το ένα πλαίσιο εδώ. Και η συνάδελφος Πιτσερίβο που εκπροσωπεί τον κύριο Δεκάστρο θα πάρει μετά το λόγο. Τώρα θα σχολιάσουμε το σχέδιο προπολογισμού για το 2020 και τα συγκεκριμένα ποσά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναλύσουμε τη θέση του Συμβουλίου που τη λάβατε από τη Γραμματεία. Φέτος, λόγω της ε, διακοπής για τι εκλογέ, η προηγούμενη Επιτροπή Άγκρη δεν έστειλε επίσημη γνώμη για την εντολή για τον ε, τριμερή διάλογο του Ιουλίου. Ωστόσο, κατέστησε σαφέ στην Επιτροπή Προπολογισμών ποια θέματα μας ενδιέφεραν μέσω επιστολής. Κατά το τέλος της ε, προηγούμενης νομοθετικής θητεία, αποφασίστηκε να ε, πάρει τη γνωμοδότηση αυτή η σοσιαλιστική ομάδα και ο κύριος Δεκάστρο ορίστηκε της λόγω του περιορισμένου χρόνου και των εκλογών. Το σχέδιο γνωμοδότηση είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. Πέρα από την τροπολόγηση αυτού του σχεδίου γνωμοδότηση που θα γίνει μέσω των ψηφοφοριών τη 4 η Σεπτεμβρίου, έχετε δυνατότητα, όπω κάθε χρόνο, να υποβάλλετε τροποποίηση του προπολογισμού για να αλλάξετε τα ποσά που προβλέπονται στο σχέδιο προπολογισμού. Υπενθυμίζω στα ε, παλιά μέλη και ενημερώνω τα νέα μέλη ότι οι πιλωτικέ δράσεις και οι προπαρασκευαστικέ ενέργειες μπορούν να γίνουν μόνο μέσω τροποποιήσεων του προπολογισμού. Αυτές οι τροποποίησεις θα ψηφιστούν παράλληλα με το σχέδιο γνωμοδότηση και θα αποσταλούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Η κυρία Πιτσέρνο. Πιτσέρνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αντικαθιστώ το συνάδελφο Ντεκάστρο, ο οποίος ε, λόγω κάποια έκτακτου γεγονότος χρειάστηκε να αποχωρήσει και μου άφησε εδώ να σας γνωστοποιήσω την άποψή του. Ο κύριος Δεκάστρο λοιπόν μου ζητά να σας πω ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος ε, της προγραμματικής περίοδου. Επομένως ο στόχος του εισηγητή ήταν να ε, εξετάσει την πρόταση προϋπολογισμού ε, διαγράφοντας όλες τις περικοπές που έχουν προβλεφθεί από το Συμβούλιο. Όχι μόνο αυτό, γιατί για κάποιους ιδιαίτερα ευαίσθητους και πολύ σημαντικούς τομές, όπως για παράδειγμα το απορροκυπευτικά, το ελαιόλαδο, το ε, μοσχαρίσιο και το βόλιο Κρέα. ζητάμε να διατηρήσουμε την παρούσα πρικοδότηση, δηλαδή του 2019, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, την ευαισθησία αυτών των αγορών. Επίσης, θα πρέπει να επενθυμίσω, κύριε Πρόεδρε, σε όλους τους ε, συναδέλφους ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες προβλέπεται για την 5η 25 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφα για αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Ο κύριος Άλβαρες τώρα, σκιώδης του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Άλβαρες πρώτος. Ο κύριος Άλβαρες πρώτος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την παρουσίαση που μας έκανε και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τεκάστρο ε, για την γνωμοδότησή του για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο δημοσιονομικό έτος, 2020. Όπως όλοι ξέρετε, δεν ήταν καθόλου εύκολο το έργο του κυρίου Τεκάστρο, γιατί ολοκληρώθηκε η προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και ξεκίνησε η καινούργια και μπράβο του, συγχαρητήρια για το αξιόλογο έργο του μέσα στο τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, ε, εσείς είστε και πρόεδρος της Επιτροπής, ε, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής, μάλλον ο κ. Τεκάσος, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, γνωρίζει ε, από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις προκλήσεις και θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες αυτές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό προϋπολογισμό που θα είναι όμως και επαρκή ταυτόχρονα για την κοινή γεωργική πολιτική που θέλουμε όλοι να προσπίσουμε. Ο σκιώδης ηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση θα κάνω προτάσεις προκειμένου να βελτιώσω την πρόταση του συντάκτη γνωμοδότης του κυρίου Παύλο Τεκάστρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και ακτινοτροφίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καντάιρα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Δεκάστρο για την ισορροπημένη του γνωμοδότηση. θα είμαι και πάλι σκιώδη και θα ήθελα να σταθώ σε μερικά σημεία. Βρισκόμαστε στην... στον τελευταίο χρόνο της προηγούμενης δημοσιονομικής περίοδου με πρόταση για πολύ ατυχή πρόταση μάλλον για αρκετές περικοπές. Λυπόμαστε για τις προτάσεις περικοπών, θα πρέπει όμως δυστυχώς να τις λάβουμε υπόψη. Σίγουρα και ο αντίκτυπος του Brexit θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, τα 50 εκατομμύρια για την Ιρλανδία, αλλά δεν θα επηρεαστεί μόνο η Ιρλανδία από τον Brexit και άλλες χώρες θα πληγούν. Η Φιλανδία και οι χώρες της Βαλτικής, για παράδειγμα, έχουν πληγεί από τις ε, ρωσικές κυρώσεις. Κάτι που εξακολουθεί να ταλανίζει τους ε, Φιλανδούς γεωργούς. Και επηρεάζει πολύ αρνητικά το γαλακτοκομικό μας κλάδο. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για τη γνωμοδότηση του κυρίου Ντεκάστρο. Καταρχήν, συμφωνώ με την παρατήρηση ότι η περικοπή του γεωργικού προπολογισμού για το 2020 είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα για το Γεωργικό Ταμείο και τα Ταμείο Αγροτικής ανάπτυξη. Προτείνεται μείωση του ταμείου αυτού κατά 13,4 εκατομμύρια ευρώ. Λυπόμαστε που η πρόταση του προπολογισμού το 2020 δεν λαμβάνει δεόντω υπόψη τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα ε, και το κεντρικό ρόλο της γεωργίας. Ε, είναι σημαντικές οι προκλήσεις ε, τη Γεωργία από τη Συμφωνία των Παρισίων. Η Γεωργία είναι θύμα των κλιματικών αλλαγών και κρίνεται και ω υπέτεια των κλιματικών αλλαγών με τα αέρια του θερμοκηπίου. Μπορεί όμω η Γεωργία να είναι και τιμά τη λύση αν την υποστηρίξουμε δεόντω για να τηρήσει τι υποσχέσει των Παρισίων για το κλίμα. Και θέλουμε η Συμφωνία των Παρισίων να ληφθεί περισσότερο υπόψη στον προπολογισμό. Θα χρειαστούν επιπλέον προσπάθειε ώστε 30% του προπολογισμού της Ένωσης ε, να, ε, να αφιερωθεί στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Επίσης, το αποθεματικό κρίσης είναι σήμερα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να στηρίζει τους πιο ευάλωτους γεωργούς, κυρίως αυτούς που έχουν πληγεί από την ε, σοβούσα ξηρασία. Όπως και ο κύριος Δεκάστρο και εγώ εκπλήσωμαι που δεν παραλείπεται τελείως το ζήτημα του Brexit. Και μάλιστα δεν λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές συνέπειες ε, της ε, αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό όμω το ανέφεραν και οι προλαλήσαντε και σα, κύριος η συνάδελφο από τη Γαλλία. Τα ερευνητικά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, του ορίζοντα 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για περισσότερη τεχνογνωσία και μελέτε για την αγροοικολογία. Κατά τη γνώμη μα, η αγροοικολογία είναι η καλύτερη δυνατή καινοτομία για να βοηθήσουμε τους γεωργούς ε, να εστεριστούν πιο θεκτικά μοντέλα για τα φυτοφάρμακα, για το κλίμα, για την διαφύλαξη της βιοπικιλότητας, αλλά και για την υγεία. Θα θέλαμε λοιπόν σημαντικά κονδύλια, πολύ υψηλότερα κονδύλια, να αφιερωθούν στην έρευνα για να παρακολουθήσουμε την ωραία αυτή καινοτομία που συνιστά η αγροοικολογία. Όλες αυτές τις πληροφορίες, όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις θα τις διαβιβάσουμε πριν τις 25 Ιουλίου, αν κατάλαβα καλά την προθεσμία, στον κύριο Δεκάστρο εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ανδριούδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον Δεκάστρο, για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο στηρίζω. Αλλά να προσθέσω κάποια θέματα. Πρώτον, αυτά τα 50 εκατομμύρια για το βόλιο αποζημίωση για τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit δηλαδή, θα τα λάβει μόνο η Ιρλανδία. Βεβαίως αυτή θα θυγεί κυρίω. αλλά και άλλες χώρες. Θα θυγούν από τη διαδικασία αποχώρηση του Ευρωπαϊκού Βασιλείου. Άρα πρέπει να αυξηθεί το ποσό για να καλυφθούν και εκείνοι. Συμφωνώ με την νόμη του συγκεκριτή, όπως είπαν και άλλοι, για την ανεπάρκεια των πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, πρέπει να δώσουμε περισσότερο στο δεύτερο, για το δεύτερο πυλώνα. Επίσης, κάτι που δεν αναφέρεται στην έκθεση, τι άλλες επιπτώσεις θα έχει το Brexit. Δυστυχώς ε, τα σημερινά νέα δεν είναι καθυσχαστικά. Δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει μέχρι το τέλος του 2020 στη χρηματοδότηση του προπολογισμού του Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα πρέπει, παρά το ότι είναι δυσχερές, να κάνουμε κάποιες ε, προβλέψεις. Πρέπει λοιπόν να επαρρυπνούμε για τα θέματα της ε, υγείας και τα φυτογενομικά Ξέρουμε ότι ο πυρετός των χείρων, η πανόλη των χείρων, έχει ελεγχθεί αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Και επίσης υπάρχουν διάφορες αιστείες της γρήπης των πουλερικών, κυρίως στην Ιταλία. Και τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία, και θα το θυμάστε κύριε Πρόεδρε, το σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε επαρκείς πόρους, να επαγρυπνούμε αν υπάρξουν τέτοια υγειονομικά προβλήματα εάν ε, προκύψουν την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούσεν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τον κύριο Ντεκάστρο για αυτήν την γνωμοδότηση. Περιέχει τα κυριότερα σημεία. Να ασχοληθώ με το 6 που είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα επαρκούς χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό είναι πραγματικά ουσιώδες. Γιατί το αναφέρω. Γιατί το Συμβούλιο στη θέση που υιοθέτησε Πρόκειται για το ε, ορίζον 2020 δηλαδή. Το Συμβούλιο λοιπόν περιέκοψε 10 εκατομμύρια. Πρέπει εμείς να εμείνουμε ότι πρέπει να τηρηθεί επαρχή χρηματοδότηση. Πρέπει να επανέλθουμε στο προηγούμενο προβλεφθέν ποσό. Και νομίζω ότι συμφωνεί και η Κομισιόν μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σταντέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την εργασία του. Να αναφερθώ στα εξή. Πρώτον, τα εξαιρετικά μέτρα τα έκτακτα μέτρα για το βόλιο στην Ιρλανδία. Πολύ καλό. Πρέπει όμως να τα συμπληρώσουμε. Συμπληρώσουμε τους πόρους για να ασχοληθούν και με άλλους τομείς και επίσης να βοηθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μπορεί να θυγούν. Δεύτερον, η σοβούσα κρίση στον τομέα της Σακάριος. Δεν έχουμε δώσει φράγκο για τον κλάδο αυτό. Προτείνω λοιπόν να υπάρξουν πιστώσεις που θα πάρουμε από αλλού, να μην αυξήσουν τον υπολογισμό δηλαδή, αλλά να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαταράξεις της αγοράς, ιδιαίτερα το άρθρο 222 του ενιαίου, της ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς. Και νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη χρηματοδότηση μια σειρά από πιλωτικά σχέδια που είναι σημαντικά για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το οποίο λείπει οι Ευρωπαίοι Γεωργοί, πιο συγκεκριμένα οι Ρουμάνοι Γεωργοί, έχουν ε, ε, χάσει πολλά, ε, έχουν υποστεί ζημίες λόγω του πανόλης των χείρων. Το θέμα είναι ότι οι ζημίες των γεωργών δεν είναι από δική τους υπετιότητα. Επομένως, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό στον προϋπολογισμό. Οι γεωργοί χρειάζονται στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Το Brexit δεν αφορά μόνο το βόλιο κρέας, ε, μπορεί να πληγούν και άλλοι τομείς. Επομένως, ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αποζημιώσεις για ζημίες ε, σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τολερέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για να επιστρέψω στον προπολογισμό, να ευχαριστήσω τον Παύλο Ντικάστρο για την γνωμοδότησή του. Έχουμε όμως μια σημαντική ανησυχία στον γεωργικό κόσμο για τις αβεβαιότητες και κυρίως για τις αβεβαιότητες στον προπολογισμό, όπως έλεγαν και οι συνάδελφοι προηγουμένω. για το Brexit. Ε, έχουμε την Βρετανική αγορά και η Βρετανική αγορά είναι ε, η πρώτη αγορά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρχει λοιπόν ένας κλάδος ε, κρέατος ε, που αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα πρέπει να υπάρχει ένας προπολογισμό παρέμβασης, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπεται για να μην προσθέσουμε και το βάρος της καθυστέρησης ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πρέπει να πω κάτι ακόμα. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα, θα κάνει στις Βρυξέλλες και πολύ ζέστη αύριο. Θα πρέπει να προβλέψουμε μηχανισμούς για αποζημίωση στις ε, ζημιές που θα υπάρξουν λόγω των κλιματικών συνεπειών. Σήμερα, για παράδειγμα, ε, όλη η Ευρώπη ανησυχεί πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε και αυτά στον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίνο. Βίνερ. Ευχαριστώ. Για το 6 καινοτομία. Τι εννοείται καινοτομία. Ελπίζω ότι κάτι θέλουμε να επιτύχουμε και για το 5. Όλα αυτά που αναφέρονται για τα παιδιά, η βιωσιμότητα είναι πολύ καλά. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ε, τα σχολικά γεύματα θα πρέπει να μαθαίνουν για τη γεωργία ήδη από τα νηπιαγωγεία. Έχω ένα ίδρυμα που ε, έχω κάνει πολλές ε, μελέτες και προσπαθώ ε, από, την, ε, από νηπιαγωγείο να μαθαίνουν να μαγειρεύουν τα παιδιά, ούτε να έχουν την αυτονομία τους. Πρέπει να τα ενισχύσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκα. Πολλοί ευρωβουλευτέ ανέφεραν ε, το πακέτο των αποζημιώσεων ε, το οποίο ανέλαβε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα στοιχήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 50 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ προτείνω οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να διαβάσει πολύ προσεκτικά τις λεπτομέρειες στο πακέτο και ποιος ε, ε, είναι ο στόχος αυτή την περίπτωση. Και αν σας ενδιαφέρει και η βιωσιμότητα θα καταρρεύσετε από το σόκο όταν θα το διαβάσετε. Διότι είναι σαφές ε, ποιος είναι ο στόχος στην η ε, Ιρλανδία, για παράδειγμα, στοχεύουν στο τομέα του βόηου ε, μικρής ηλικίας. Ε, τους ενδιαφέρουν να καταστρέψουν τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Αναφέρονται ε, στο στον πιο βιώσιμο τομέας, τομέα του βόηου γάλακτος, αλλά αγνοούν τους άλλους τομείς. Αν πραγματικά λοιπόν θέλετε να δείτε πώς δαπανούνται καλά τα χρήματα, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, θα πρέπει να εξετάσετε πολύ προσεκτικά αυτό το έγγραφο. Διότι αυτό το οποίο προσφέθηκε στην Ιρλανδία δόθηκε επί της βάσης ότι οι πιο βιώσιμοι ε, κτηνοτρόφοι βόηου κρέατος θα φύγουν και θα φύγουν από τη μέση για το κρέας από τη Μερκοσούρ. Ε, δίνουμε χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου για να φύγουν από τη βιώσιμη παραγωγή ε, Περιμένο Περιμένω ε, να το θέσει αυτό η Επιτροπή Διοντολογίας. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Δεσόκλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι λόγω και των διαφόρων ανταλλαγών απόψεων που είχαμε με τον Επίτροπο και τα όσα ακούσαμε εδώ από τους συναδέλφους, οι γεωργοί έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε. Και νομίζω ότι σήμερα με όλα τα μηνύματα για τη Μερκοσούρ, ε, την ανησυχία για την ξηρασία, την ανησυχία για το βόιο, για τη ζάχαρη, αλλά και άλλους τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν ίσως να ε, πληγούν από διάφορα θέματα, σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει να βρούμε ε, επιχειρήματα για να πούμε ότι η πτώση του προπολογισμού ή η μείωση της χρηματοδότησης για τους γεωργούς δεν είναι αποδεκτή. Ακόμα κι αν ε, όπως διαπιστώνουμε όλοι, πρέπει να δώσουμε μάχη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ε, μόλις επιβεβαίωσε και τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ και να τους πούμε ότι κάποια στιγμή δεν μπορούμε να ε, βάζουμε εμπόδια στους γεωργούς και στη γεωργία και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουμε και το ρίσκο να διαπραγματευόμαστε τέτοιες συμφωνίες, διότι δίνουμε τελείως λανθασμένα ε, μηνύματα στους γεωργούς και φυσικά ε, δεν τους δίνουμε κίνητρα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του κλίματος, αλλά και άλλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Ευχαριστώ η κυρία... Μπορείτε να συνοψίσετε. Ναι, αλλά μόνο όταν τελείωσαν οι παρεμβάσει όλων των συναδέλφων. Τελείωσαν, ωραία. Κυρία Πιτσέρνο. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω όλου εξ ονόματο του συναδέλφου Ντεκάστρο για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε και τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις τους και ε, θεωρώ ότι θα βρεθεί τρόπος να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο όπου θεωρείται ότι πρέπει να προσθεθούν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και να υπενθυμίσω όπως είπα και στην αρχή ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η 25 Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για αυτή την γνωμοδότηση και για τη συζήτηση. Θα εγκριθεί στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας. Στην ε, Επιτροπή ε, Αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμών δηλαδή ή θα είναι τη βδομάδα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Οπότε τώρα, να περάσουμε... Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο, με συγχωρείτε. Ναι, επειδή ετέθησαν μερικά ερωτήματα. Αν θέλετε να απαντήσω, αλλά όπως θέλετε. Α, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Αλλά επειδή ετέθησαν ορισμένα θέματα που μπορούμε να διευκρινίσουμε και μάλλον θα έπρεπε πριν ε, διαμορφώσετε την τελική σας άποψη για αυτά. Πρώτον, διάφοροι ευρωβουλευτές είπαν ότι γίνονται περικοπές για την ανάπτυξη της πέθρου. Δεν υπάρχει καμία περικοπή για την ανάπτυξη της πέθρου, να το διευκρινίσουμε. Υπάρχει μια ελαφρά μείωση 13 εκατομμυρίων αλλά είναι μόνο τεχνική βοήθεια. Δεν είναι πόροι για τα προγράμματα ή για να βοηθηθούν οι παραγωγοί. Είναι κυρίω το διοικητικό κόστο των κρατών μελών, το οποίο μειώθηκε. Να διευκρινίσω. Δεν υπάρχει καμία μείωση των πόρων για την ανάπτυξη τη υπαίθρου στο σχέδιο προπολογισμού του 2020. Για τον Brexit. Λοιπόν, και εδώ σου χρειάζονται κάποιε διευκρινήσει. Ο προπολογισμό βασίζεται στην συμμετοχή τη χρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση και των 28 με βάση τη συμφωνία αποχώρηση του Ηνωμένου Τώρα μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει κίνδυνο ότι δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Αλλά όταν προτάθηκε αυτό ο προπολογισμό, ήμασταν υποχρεωμένοι να βασιστούμε στα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο έκανε μια ανακοίνωση, την οποία επιβεβαίωσε μέσω άλλη ανακοίνωση τον Ιούνιο για την ε, προπαρασκευή για τον Brexit, όπου λέγεται σαφώς ότι εάν για κάποιους τομείς, ιδιαίτερα στη Γεωργία, υπάρξουν ε, διαταραχές της αγοράς, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη, είναι έτοιμη να κάνει πρόταση οικονομικής ενίσχυσης. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ε, αυτό συμβεί στις 31 Οκτωβρίου θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Για το πακέτο βοήθειας προς την Ιρλανδία. Έχουμε το παρατηρητήριο αγορών, μέσω του οποίου παρατηρούμε τι γίνεται σε όλες τις ε, αγορές γεωργικών προϊόντων, όχι μόνο για το Βόρειο, όχι μόνο στην Ιρλανδία. Και με βάση την ενημέρωση που έχουμε, διατυπώσαμε αυτή την πρόταση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που προέκυψε στην Ιρλανδία. Αλλά εάν ε, υπάρξει κάτι άλλο στι αγορέ και πάλι είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί. για την ε, γρήπη των πουλερικών στην Ιταλία. Το σχέδιο προπολογισμού δεν είναι ενημερωμένο γιατί υπήρξε μια συνεδρίαση τη Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα που πρότεινε συγκεκριμένη στήριξη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ε, γρήπη των πουλερικών στην Ιταλία. Θα μπει κατόπιν μέσω τη διαδικασία συνδιαλλαγή. Θα είναι μήμα τη διαδικασία συνδιαλλαγή για τον προβλησμό του 2020 για την Αφρική, Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στη Ρουμανία. Εάν υπάρξει συγκεκριμένο αίτημα από πλευρά ενό κράτου μέλου για να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, είμαστε διατεθειμένοι να δράσουμε όπω και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα στην περίπτωση τη Ρουμανία. Αλλά δεν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα από τη Ρουμανία για αυτό το θέμα. Άρα δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με το θέμα αυτό ο προπολογισμό του 2020. Τέλος, για τα πιλωτικά προγράμματα. Είχαμε μία πρώτη αξιολόγηση και τώρα στο δεύτερο γύρο αξιολογούμε όλες τις προτάσεις που έχουμε που θα είναι τμήμα της συζήτησης μαζί σας αργότερα όταν θα οριστικοποιηθεί ο προπολογισμό του 2020. Και ακόμη πιο τελευταίο, για τα οποροκυπευτικά όπως λέει και ο εισηγητής, εκφράζει την απογοήτευσή του για τη μείωση, για την περικοπή. Όχι. Με βάση τις ενημερώσεις που πήραμε τα κράτη-μέλη, όλα τα αιτήματα που επιβλήθησαν, τα ικανοποιεί ο προπολογισμό αυτό, το σχέδιο προπολογισμού. Να καταστεί σαφέ, δεν υπάρχει περικοπή. Και ακόμη πιο τελευταίο. Κυρία Τολγαέ, η επίπτωση του κλίματος ε, στη Γεωργία. Αυτό δεν είναι θέμα του προϋπολογισμού του 2020. Είναι θέμα της διαπραγμάτευσης για το επομενο πολιτέ πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις επεξηγήσεις, πολύ χρήσιμες, για την οριστικοποίηση της γνωμοδότησής μας. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Άγκρι. Τα έχετε λάβει. Λοιπόν, αύριο, αν δεν έχουν υποβληθεί παρατηρήσεις, εγκρίνονται. Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς. Όχι, και ήδη τώρα. Εγκρίνεται. Σημείο 9. Διάφορα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Ούτε εσείς. Ωραία. 10. Επόμενη συνεδρίαση. 4 Σεπτεμβρίου, 9 με 12.30 και 14 με 6.30 και 9 με 12.30 στις 5 στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό βράδυ, καλές διακοπές και σας εύχομαι να επιστρέψετε υγιείς την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πέρασε.